Meine Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen und auch ruhig zu sein auf den billigen Plätzen. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Παρακαλώ για ησυχία στην αίθουσα. Χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω ε, έναν αριθμό εθνικών βουλευτών. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία στην πράξη, οι διαβουλεύσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών στα διάφορα επίπεδα, από μεγάλες διασκέψεις μέχρι εδώ στο δικό μας επίπεδο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα υπόλοιπα θεσμικά οργανά, συζητούμε για την ε, επανεξέταση της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Και είναι καλή η στιγμή για να προβληματιστούμε σχετικά με τις ελλείψεις μας. Είναι σαφές. Και την τρίτη στην Επιτροπή είπαμε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ακόμη δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη. Υπάρχουν ελλείψεις, διότι μέσα σε δύο χρόνια δεν μπορούμε να τελειοποιήσουμε μια τέτοιου είδους υπηρεσία. Υπάρχουν ε, και θέματα συνθήκης, θέματα ε, διαρθρωτικά, ε, θέματα δομής των φορέων λήψης αποφάσεων, όλα αυτά χρήζουν ακόμη βελτιώσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που με τους Υπουργούς Εξωτερικών Μπίλτ και Σικόρσκι μπορούμε να μιλήσουμε για την ε, νέα Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική, European Global Strategy, διότι εδώ χρειάζεται μια συλλογικότητα και μια συλλογική προσέγγιση για καλύτερα αποτελέσματα. Μια τέτοια συλλογική προσέγγιση θα μας βοηθήσει στο μέλλον μπορεί να έχουμε λιγότερες στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, αλλά θα έχουμε μια ενιαία στρατηγική κοινή η οποία μας λείπει και θα έχουμε και μια χρειαζόμαστε μια μέθοδο, ένα μηχανισμό για να καταλήξουμε εκεί και να μπορέσουμε να ε, συμβιβάσουμε τις ανάγκες μας με την οικονομική κρίση και τους οικονομικούς περιορισμούς λαμβάνοντας υπόψη την γεωπολιτική θέση της Ένωσης και τα γεωπολιτικά μας ε, συμφέροντα ε, λαμβάνοντας ε, παράλληλα υπόψη και προάγοντας τις δημοκρατικές μας αξίες και πρότυπα. Θα ακούσουμε τους δύο υπουργούς των εξωτερικών ε, για 15 λεπτά ο καθένας και μετά θα παρέμβει και ο δόκτωρ Αντώνιο Μισιρόλη, ο οποίος είναι διευθυντής ε, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Μελετών για την Ασφάλεια. Και θα ακούσουμε και ορισμένες εισαγωγικές παρατηρήσεις από τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, ΣΕΝΤΕ. Σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσία σας κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όπως σας υπενθύμισε ο Πρόεδρος, το 2013 είναι έτος ασφάλειας άμυνας και προσφέρει διάφορες δυνατότητες αυτή η χρονιά, διότι υπάρχει μια ιδιαίτερη όθηση που δίδεται από τις δράσεις της, υπηρεσία της υπηρεσίας και είναι ένα θέμα η ασφάλεια και η άμυνα που συμπεριέλαβε και το ε, Συμβούλιο στην ε, ατζέντα του. Υπάρχει το Ειδικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν ε, θετικές εξελίξεις. Βλέπουμε την κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ. Βλέπουμε πόσες δυνατότητες έχουμε για να βελτιώσουμε την κοινή μας ανταπόκριση, το συντονισμό μας, για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές τις οποίες δεν μπορεί κανένας μόνος του να αντιμετωπίσει παρά τις αυταπάτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και παρά το γεγονό ότι σήμερα οι Γάλλοι έχουν επιτυχία στην στρατιωτική επιχείρηση στο Μαλί. Πιστεύω όμως ότι τελικά κανένας δεν θα μπορέσει μόνος του να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις απειλές οι οποίες γίνονται στις γειτονικέ μας περιοχές, η Ανατολικά ή Νοτίως. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο να υπάρξουν πρωτοβουλίες όπως αυτές που θα μας εξηγήσουν σήμερα προσκεκλημένου, ώστε να μπορέσει να κάνει αιρέση των προτεραιοτήτων τη και ορισμό των προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι χωρί να ορίσουμε τι προτεραιότητε, θα κάνουμε οτιδήποτε, αλλά όχι το σωστό ενδεχομένω. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να ταυτοποιήσουμε τι απειλέ και τι προκλήσει για να δούμε πώ θα τι αντιμετωπίσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε οι εραχόντες τη. Γι' αυτό πρέπει να πω ότι είμαστε θετικοί προς τις ε, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται. Είναι πολύ θετικά αυτά τα think tank τα οποία έχουν ε, ε, δημιουργηθεί και ελπίζω ότι με αυτά τα οποία θα ακούσουμε, με αυτά τα οποία έχει αναλάβει και ο κύριος Καλμπίλτ μεταξύ των άλλων, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ. I continue in English, I can assure you. <laughs> Um, Μπορώ να σα διαβεβαιώσω. Ευχαριστώ για την πρωτοβουλία. Με ευχαρίστηση πάντα έρχομαι στην Επιτροπή σα και πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία το ότι καλέσατε στι συζητήσει σα και καλείτε που και που εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ωραία μέρα σήμερα. Φαίνεται ότι είναι κάπως καλύτερα σήμερα σφαιρικά η Ευρώπη από ό,τι πριν από μερικούς μήνες παρά το γεγονό ότι υπάρχει μια κάποια σύγχυση, δεν είναι καταστροφική κατάσταση. Πλησιάζουμε το 2014, έτος κατά το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα για το τι ακριβώς έγινε τον προηγούμενο αιώνα και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της Ευρώπης και για το μέλλον του κόσμου. Τον Ιανουάριο και τον ε, Φεβρουάριο ε, πριν από 20 ε, χρόνια πριν το 1993 υπήρχε ο Πόλεμο στη Βοσνία, άλλα προβλήματα, αλλά η οικονομία καλά τα πήγαινα. Και στη Βιέννη υπήρχαν δύο νέοι άνθρωποι που περπατούσαν κάθε πρωί, από όσων ξέρουμε. Ένας από αυτούς ήταν, συγγνώμη, το 1913 ο Αδόλφο Χίτλερ. Και δεν ξέραμε τι θα κάνει ε, σε αυτόν τον κόσμο τον αιώνα του. Ο άλλος ήταν στην ε, Βιέννη για δύο εβδομάδες ο Στάλιν. Δεν ξέραμε και αυτός θα κάνει τον Ισραήλ. Πού να ξέραμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έκαναν αυτό που έκαναν και οι δύο στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η αρχή μιας ε, καταστροφής, η οποία κατέστρεψε την Ευρώπη και υπονόμευσε και τη μοίρα του υπόλοιπου κόσμου κατά κάποιο τρόπο. Τα 20 τελευταία χρόνια είδαμε πόσες αλλαγές έγιναν στην Ευρώπη και τι προσπάθειες έγιναν να αποκατασταθούν ε, οι καταστροφές που άρχισαν το 1913 και μετά. Το 2014 μια πολύ σημαντική χρονιά, νέα χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευρωπαϊκές ευρωεκλογές. Ο Έλμαρ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι θα γίνει και αναθεώρηση των μέσων τα οποία δημιουργήθηκαν για να μπορέσει να δημιουργηθεί η, Ευρω... εξωτερική... η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέσα που ακολουθούν, ποιε είναι οι δράσει που ελήφθησαν και πώ θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε όλα αυτά ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γίνει αναθεώρηση του hardware λοιπόν των ε, Ευρωπαϊκών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρώμη δεν έγινε όπως λέμε σε μία μέρα. Το ίδιο δεν μπορεί να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι αναθεωρώντας το hardware θα πρέπει να δούμε τι κάνει και το software, το λογισμικό. Το ένα χωρίς το άλλο δεν μπορεί να δουλέψει και μπορεί να είναι άχρηστο το λογισμικό αν δεν υποστηρίζεται από το hardware και ε, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το software των πολιτικών που ακολουθούμε και θέλουμε να εφαρμόσουμε. Έχουμε την ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική, Σφαιρική Στρατηγική 2013. Πρόκειται για ένα πολύ καλό έγγραφο, έγγραφο το οποίο δημιουργήθηκε μεσούσης μια πολύ μεγάλη κρίση των διατλαντικών σχέσεων και ασχολήθηκε με τα βασικά της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό το έγγραφο ήταν εκείνη την εποχή προευρωπαϊκό, ενώ υπήρχε η αντίθεση αυτών που έκανε η κυβέρνηση Μπούς. Ε, εκείνοι μιλούσαν για μονομερή ανταπόκριση, εμείς για πολυμερή. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι μία δεκαετία αργότερα πιο πολλά έγκυρα σημεία υπάρχουν στο δικό μας έγγραφο για το μέλλον, παρότι στο αντίστοιχο έγγραφο των Αμερικανών για το μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι μαρτυρία της ε, ενόρασης που είχαν οι Ευρωπαίοι για το μέλλον και την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε μια νέα κατάσταση. Το έγγραφο αυτό ε, έγινε, εκτυπώθηκε πριν από την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνης και την ε, τελευταία διαβρύνση. Τότε είμαστε 15 μέλη. Πέρασαν χρόνια από τότε. Και ο κόσμος όντως άλλαξε και αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης άρχισε σε ένα κόσμο ο οποίος είχε γύρω στα 2,5 δις, γιατί σήμερα έχουμε 7 δις. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με τις προβλέψεις βαδίζουμε προς τα 9 δις και εμείς οι Ευρωπαίοι θα είμαστε σε λίγα χρόνια σε αυτό το νέο κόσμο το 7%. 9% της οικονομικής ε, παγκόσμιας ανάπτυξης, δεδομένου ότι θα ανακτήσουν μια πολύ καλή ταχύτητα οι άλλες χώρες. Καλό είναι αυτό, διότι σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν λιγότερες διαφορές, υπάρχουν ε, αναδυόμενες νέες οικονομίες, αλλά και νέες προκλήσεις και αντιθέτεις. Έτσι λοιπόν άρχισε πριν από μερικά χρόνια η νέα φάση, μια πρώτη φάση ε, παγκοσμιοποίησης, άρχισε η δεύτερη όπως ξέρουμε και αυτή τη στιγμή είμαστε στην τρίτη που είναι η επάνωδος της Κίνας, των Ιαπώνων, των Ινδών, των Ιαπωνέζων, για να μπορέσουν να ανακτήσουν την ε, ε, θέση που είχαν στον κόσμο πριν από δύο αιώνες. Και αρχίζουμε ίσως να βλέπουμε και τα πρώτα μηνύματα της ε, ενίσχυσης και της Αφρικής. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Προκλήσεις για μας τους Ευρωπαίους. Προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Και αν δούμε πραγματικά τι θέλουν οι εκλογείς μας να κάνουμε, το ως ορισμένοι ή εκλεγμένοι ε, υπεύθυνοι των κρατών μελών μας, πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, να μην έχουμε τόσο ε, αντίθετες και ε, ε, ιδεολογίες σε αντιπαράθεση, να μην έχουμε τα προβλήματα ταυτότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα βλέπουμε να είναι πιο έντονα, όλο και πιο έντονα στον Ισλαμικό κόσμο, που είναι οι εγκύτεροι γειτονέ μας, όχι μόνο βλέποντας το γεωγραφικό χάρτη, αλλά βλέποντας και τον κόσμο στον οποίο ζούμε, τις χώρες μας και τις διάφορες οικίες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αμβλύνουμε όλα αυτά τα προβλήματα, να λύσουμε καλύτερα. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι όλο και περισσότερο ε, συνδεδεμένος ε, μεταξύ του και επικοινωνεί όλο και περισσότερο. 85% 100 ε, ε, του κόσμου σε μερικά χρόνια θα είναι συνδεδεμένος με, την, ε, με τα μέσα κινητής ε, τηλεφωνίας ευρυζωνικά. Το βλέπουμε αυτό παντού, σε όλες τις ε, υπήρους και αυτό δημιουργεί νέες δυνατότητες. Άρα ε, μας επηρεάζει όχι μόνο ότι γίνεται γεωγραφικά αν θέλετε, αν δούμε το χάρτη της οικουμένης σε αυτή την περιοχή στην άλλη περιοχή, αλλά βλέπουμε τι ακριβώς στον σημερινό κόσμο συμβαίνει ε, στον οικονομικό τομέα, με τις επενδύσεις, τα κεφάλαια, την καινοτομία, το εμπόριο και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα θέματα επηρεάζουν τον κόσμο, επηρεάζουν την ισορροπία δυνάμεων, την αλογία δυνάμεων. Βλέπουμε τι συμβαίνει και στο διάστημα. Βλέπουμε τι συμβαίνει στον ε, κυβέρνοχώρο. χώρο. Συνειδητοποιούμε ως τι γίνεται. Επίσης, ε, πάντα ε, στο διάστημα στον κυβερνοχώρο έχουμε τις κατάλληλες πολιτικές, έχουμε τα καλά τα μέτρα και εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να αντιποκριθούμε στις προκλήσεις και να επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω τις προκλήσεις οι οποίες θα έχουμε μπροστά μας εξαιτίας κλιματικής αλλαγής που είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτές τις μέρες στο Συμβούλιο είδαμε τι γίνεται στην ε, περιοχή της ε, Αρκτικής. Δεν είναι τόσο μακριά. Βλέπουμε ε, ότι θα δημιουργηθεί μια νέα γεωστρατηγική ε, περιοχή που θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε όλους τους τομείς πριν να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα και είναι πάρα πολύ αργά. Τα αναφέρω όλα αυτά, διότι πρόκειται για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Το έγγραφο λοιπόν του 2003 ήταν πολύ καλό, αλλά τα πράγματα αλλάζουν, είναι μεγαλύτερη, πιο φιλόδοξη, πιο ισχυρή η Ευρώπη, αλλά υπάρχουν σήμερα πολλές περισσότερες και διαφορετικές προκλήσεις από το 2003. Ο Υπουργό Κόσκι και άλλοι, όπως και εγώ, προσπαθήσαμε να κάνουμε μία πιο διεξοδική ε, και επικυρωμένη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι πώς θα μπορέσουμε με στρατηγικές επιλογές και μέσα να αλλάξουμε τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι για να μπορέσουμε να ξέρουμε τι γίνεται και εκτός ε, ε, των ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων δημιουργήσαμε τέσσερα think tanks στην Ιταλία, στην Πολωνία, την Ισπανία και τη Σουηδία για να ακούσουμε τις φωνές όλων και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και θα μου πείτε τι περίεργο συνδυασμός χορός είναι αυτός. Ακούστε. Είναι αρκετά ευφιές το όλο σύστημα έτσι όπως οργανώθηκε ή τουλάχιστον αυτό σκεφτόμαστε. Πρόκειται για χώρες από το βορρά, από το νότο, μία χώρα που ήταν από τις πρώτες που ε, δημιούργησαν την Ευρώπη, από την Ανατολή, από τη Δύση, από τον Βορρά και βεβαίως δεν είναι όλες απαραίτητος από τις μεγαλύτερες. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ ευφύ συνδυασμό χωρών και think tanks. Θα δούμε ποιο θα είναι το έργο που θα παράξουν. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι ανοιχτή σε όλους. Διότι σε τέτοιου είδους ε, διαδικασίες πρέπει να πούμε ότι τόσο η διαδικασία όσο και το προϊόν που θα παράξουν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα έγγραφο 10, 15, 20, 25 σελίδων κάποια στιγμή θα το φτιάξουν και ίσω θα δεμόσουν, αλλά είναι σημαντικό το περιεχόμενο και σημαντικό τρόπο τον οποίο όλοι θα μελετήσουν και θα σκεφτούν στις χώρες μας για να μπορέσει να γίνει τελικά αυτό το έγγραφο. Και όλη αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική διότι θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας κάποια συνένεσης στην οποία θα καταλήξουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική. Αυτά λοιπόν σε γενική γραμμές είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις πολύ μεγάλες αλλαγές οι οποίες θα συμβούν. Δεν είμαστε στο 1913, ε, αλλά νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι πολύ περισσότερες από όσο μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι ότι υπάρχουν προκλήσεις υπάρχουν δυνατότητες και το καθήκον μας είναι να εφαρμόσουμε τη σωστή στρατηγική και τελικά να διαμορφώσουμε τα μέσα, τα εργαλεία και τις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω τη συζήτηση αυτή, δεδομένου ότι είναι μέρος της όλης αυτής της διαδικασίας, την οποία ελπίζω θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα επόμενα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε στα πλαίσια αυτής της ευρωπαϊκής συνολικής στρατηγικής να έχουμε τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό που θα μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές και τις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός Σικόρσκι. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ. Την τελευταία φορά είχα τη χαρά και την τιμή να σας απευθύνω το λόγο όταν παρουσίασα τις προτεραιότητες της Απολωνικής Προεδρίας το 2011. Και τότε ανησυχούσα για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Τώρα ανησυχώ για μια Ευρώπη χωρίς ταχύτητα. Το πρόβλημα του να παίρνει κανείς το λόγο μετά από έναν έγκυρο μιλητή όπως ο Καρλ Μπίλτ είναι ότι συμφωνεί με όλα όσα είπε. Συνεργαζόμεθα τόσο στενά που είναι συγχρονισμένες σχεδόν οι απόψεις μας. Είμαστε στη Μολδαβία τις προάλλες με τον Βίλιαμ Hague μαζί προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους Μολδαβούς στην πολιτική τους διαδικασία και τις διαπραγματεύσεις για να επιτύχουν συμφωνία σύνδεσης μαζί μας. Θες στο Ντάνσκ υπήρξε νέα πρωτοβουλία της πολωνικής κυβέρνησης και της ομάδας Βίσεγκραντ, γιατί η ομάδα Βίσεγκραντ και το ε, Συμβουλίο Βορείων Χωρών και των Σκανδιναβικών Χωρών ανέλαβαν πρωτοβουλία και στις Βρυξέλλες και στην Βαρσοβία. Ε, στη Βαρσοβία παίρνω το λιγότερο χρόνο. Ε, βλέπω πιο πολύ τους συναδέλφους παρά την οικογένειά μου. Θα μπορούσα να προσθέσω κάποια επιχειρήματα σε αυτά που παρέθεσε ο Υπουργό σχετικά με το πώς θα διαχειριστούμε τη θέση της Ευρώπης σε έναν κόσμο στον οποίο δεν είμαστε η κυρίαρχη πλέον ε, οικονομική και δημογραφική δύναμη. Η Ευρώπη πρέπει να πούμε ότι αρκετά καλά τα πήγε δεδομένης ε, της κρίσης, με καθαρά οικονομικά κριτήρια μιλώντας. Ε, έχουμε κάποια στοιχεία. Το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία ήταν σταθερό στο 20% την πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα. Το μερίδιο των ΙΠΑ μειώθηκε κατά 12% και της Ιαπωνίας κατά 5%. Οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι η μείωση είναι σχετική. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η μείωση είναι σχετική, αλλά αυτά είναι τα στοιχεία. Με την κακοδιαχείριση της χρήσης ε, μειώσαμε το κύρος μας στον κόσμο. Και αυτό είναι μέρος του συσχετισμού δυνάμεων. Αυτή είναι μια ορολογία ε, από τη Σοβιετική εποχή, αλλά χρήσιμη εδώ. Τώρα υπάρχει το επιχείρημα ότι εμείς αν συνενώσουμε τις ε, δυνάμεις μας θα είμαστε ισχυρότεροι. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Χάρολτ Μακμίλαν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός παλαιότερα είπε και παραθέτω ότι η Ευρώπη είναι στην θέση των ε, ελληνικών ε, πόλεων εθνών αντιπάλεψαν, πολέμησαν το ένα το άλλο και κατέρευσαν. Ε, πρώτα κυριάρχησε ο Μέγας Αλέξανδρος, μετά οι Ρωμαίοι, η Ευρώπη ενωμένη θα μπορούσε χωρίς να κάνει παζάρια για το μέγεθος των φορτηγών, αλλά με μια ενιαία εξωτερική πολιτική, μια ενιαία αμυντική πολιτική και μια οικονομική πολιτική θα μπορούσε να εξισωθεί με τις μεγάλες υπερδυνάμεις. Το επιχείρημα του Μακμίλαν εξακολουθεί να είναι σωστό, αλλά η πρόκληση ε, εξακολουθεί να είναι το ίδιο μεγάλη. Εξακολουθούμε ε, να ε, αντιτιθέμεθα ένα στον άλλον. Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Μιλήσαμε για κοινή στρατηγική, για κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική εξωτερικής δράσης, αλλά πολλά κράτη-μέλη μπαίνουν στον πειρασμό να δράσουν μόνα σε σχέση με κάποιους στρατηγικούς εταίρους στην Ευρώπη, της Ευρώπης αν κάνουμε μια προβολή των τωρινών τάσεων στο μέλλον. Και αν είναι αλήθεια ότι ακόμα και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις νέες εξελίξεις. Ε, για παράδειγμα, το μερίδιο της ε, Γερμανίας φαίνεται ότι από το τωρινό 4% θα πέσει στο 2%. Σε λιγότερο από 50 χρόνια η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, οι τρεις μεγάλοι, ε, θα έχουν ένα μερίδιο μόνο 6% και οι τρεις μαζί, δηλαδή το μισό από το τωρινό μεριδιό τους. Φαίνεται ότι το 2050 καμιά ευρωπαϊκή, εθνική ενώ οικονομία δεν θα συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων παγκόσμιων οικονομιών. Οπότε το επιχείρημα υπέρ της συνεργασίας ε, των 500 εκατομμυρίων που συλλογικά έχουν το 25% συνολικά του παγκοσμίου ΑΕΠ, είναι ένα ισχυρό επιχείρημα. Τώρα το θέμα είναι μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Ο Κάρλ μίλησε για το software, για το λογισμικό. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Νομίζω ότι το hardware που έχουμε δεν ε, μας το επιτρέπει αυτό. Δεν είναι προσανατολισμένο προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσωπικά πιστεύω ότι η ύπατη εκπρόσωπος, για παράδειγμα, ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε στο μέλλον να τεθεί επικεφαλής ενός κλάστερ, μιας συσπήρωσης αν θέλετε, μιας ομάδας επιτρόπων, ούτως ώστε να μπορεί να αναπτύσσει τα μέσα και τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που έχουμε. Αυτό δεν είναι μόνο διπλωματία. Είναι διπλωματία η οποία στηρίζεται, δράζεται σε πόρους που είναι αναπτυξιακοί, γιατί ε, είμαστε ε, ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός εταίρος στον κόσμο και ίσως μια άλλη συσπήρωση ομάδα που θα στηρίζει τη διπλωματία μας με πιθανή χρήση ε, άσκησης δύναμης, ισχύως. Πέρσι η κάθε Άστον ε, έδωσε τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιούν ε, όπλα κατά των εχθρών, των πειρατών στις ακτές της Σομαλίας. Αυτό έγινε και με μεγάλη επιτυχία μάλιστα. Το ποσοστό πειρατεία σημειώθηκε κατά 70%. Ε, Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία που οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν τη γνωρίζουν. Και εδώ θα διαφοροποιήσω λίγο τις προτεραιότητες από τον Καρλ, γιατί νομίζω ότι για να είναι κανείς αποτελεσματικός στον παγκόσμιο καταμερισμό δυνάμεων και για να είναι κανείς σεβαστός και στην Κίνα και στη Βραζιλία και στην Ουάσιγκτον και παντού, πρώτα απ' όλα είναι να τακτοποιήσουμε τα της γειτονίας μας. Εκεί ασκούμε και τη μεγαλύτερη επιρροή. Εκεί οι πόροι μας Ε, επηρεάζουν τους γείτονες και τους πείθουν να συνεργαστούν μαζί μας και εκεί είναι ε, πιο εύκολη η πολιτική μας. Αν αποτύχουμε στην άμεση γειτονική μας περιοχή θα αποτύχουμε και αλλού. Νομίζω λοιπόν ότι το έτος των ε, θεμελιωδών αποφάσεων δεν είναι κατά το παρελθόν όταν δημιουργήθηκε η Ένωση, αλλά φέτος, γιατί φέτος ε, ο, θα αποφασιστεί ο γεωπολιτικός προσανατολισμός των ε, εξανατολών γειτόνων μας. Στο Νότο έχουμε γείτονες της Ευρώπης, στην Ανατολή έχουμε Ευρωπαίους εταίρους, κάποιες χώρες έχουν ω όραμα να αποκαταστήσουν πολύ πιο στενέ σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέτος θα γίνει σύνοδος κορυφής στο Βίλνιου τη ανατολική εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η ανατολική εταιρική σχέση θα μπορούσε να είναι σύνοδος κορυφής που θα σηματοδοτήσει νέα αρχή της εταιρική σχέσης προς Ανατολάς και θα μπορούσε επίσης να ε, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ε, θα μπορούσα να φανταστώ στη Σύνοδο Κορυφή των ε, Νοέμβριων η Ουκρανία να υπογράψει συμφωνία σύνδεσης και μέχρι και τρεις από τους ανατολικούς γείτονες να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις και ίσως να μονογραφήσουν και συμφωνίες σύνδεσης. Μια νέα μορφή συμφωνία, συμφωνιών σύνδεσης με ε, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών μεγάλες και έτσι θα αναλάβουν τη δέσμευση να υλοποιήσουν το 60% του, του ενωσιακού κεκτημένου στο δικαιικό του σύστημα. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη για την επιτυχία του Βίλνιους. Γνωρίζετε όμως εξίσου καλά όπως και εγώ ότι η εναλλακτική σε αυτό είναι οι χώρες αυτές να προσανατολισμούν να προσανατολιστούν συγγνώμη, προς μια ε, διαδικασία ολοκλήρωσης ε, ανταγωνιστική που δεν θα επικεντρώνεται σε μας, αλλά θα, θα ε, προσεγγίζει άλλα φιλόδοξα σχέδια ολοκλήρωσης. Έτσι λοιπόν πρέπει να δώσουμε την προτίμησή μας εδώ, γιατί αν ξέρουμε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει την ισχύ να προσελκύει άλλους, ότι εξακολουθεί να αποτελεί κάτι στο οποίο προσβλέπουν άλλοι, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποιο ε, χαμένο έδαφος. Εγώ είμαι πρώην Υπουργός Άμυνας ο προηγούμενος ε, άλλοι ήταν ε, Τα μαθήματα που άντλησα από τις ε, επανεξετάσεις μας και τις στρατηγικές που έχουν πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι δεν πρόκειται για θεωρητικά έγγραφα. Στον τομέα της άμυνας ε, κάποιες επανεξετάσεις που έχουν νόημα αφορούν τις δαπάνες. Αυτό που η στρατηγική ελπίζω να μας εξοπλίσει για να κάνουμε δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε μια συνένεση γύρω από τις πολιτικές μας, αλλά μια συνένεση και γύρω από τις δαπάνες. Συχνά υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ των λεγόμενων και των γραφωμένων μας και των πραγματικών δαπανών μας. Ελπίζω λοιπόν ότι η στρατηγική αυτή θα δημιουργήσει συνένεση στην δημιουργία νέων hardware, νέων μέσων και θα μπορέσει να ε, συνδυάσει τις φιλοδοξίες μας και την ιεράρχησή μας και στον τομέα των δαπανών. Αν πούμε ότι η Βόρεια Αφρική αποτελεί προτεραιότητα ε, δηλαδή είναι σημαντική για τη σταθεροποίηση των γειτόνων μας και ισχύει αυτό γιατί εκεί υπάρχει η κρίση, αυτό πρέπει και να αντικατοπτρίζεται στον επιμερισμό των πόρων μας, των κονδυλίων μας, λυπούμε που θα το πω, σε βάρος άλλων περιφερειών. Πρέπει να γίνει αυτό. Σίγουρα αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα, γιατί για ιστορικούς λόγους κάποια κράτη-μέλη μας ε, θεωρούν ότι έχουν ιστορικές ευθύνες για κάποιες περιοχές. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Αν δεν συνδυάσουμε τις δαπάνες μας με τις δεδηλωμένες πολιτικές μας, δεν θα επιτύχουμε πολλά. Θα μείνουμε στα παραδοσιακά. Ελπίζω ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και νομίζω ότι έχουμε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι ότι θα μπορέσει η στρατηγική μας να είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μισηρόλη. Uh, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να από αποτανθώ σε εσάς σήμερα μαζί με τους ε, Υπουργούς Εξωτερικών. Θα ήθελα να σας πω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ασχοληθεί με μια στρατηγική εξωτερικής πολιτικής γενικότερα. Θα ήθελα να πω ότι αν δούμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τα τελευταία 20-30 χρόνια, οι πιο επιτυχείς στρατηγικές ε, που ακολουθήσαμε σπάνια είχαν παρουσιαστεί ως επιτυχείς στρατηγικές. Δηλαδή, η διεύρυνση προήλθε από ένα πολύ περιορισμένο άρθρο της συνθήκης. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Σέγγεν ήταν ε, μία διαδικασία επέκτασης από ένα μικρό πυρήνα. Όλες οι ιστορίες επιτυχίας είχαν ε, μεγάλη επίπτωση στην εξωτερική μας πολιτική και βοήθησαν ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι δελεαστική για αυτό που είναι και για αυτό που πράττει ή αναφέρει. Επρόκειτο για μέσα, για μια εξωτερική πολιτική μέσω άλλων πολιτικών. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος αφορά ένα γενικότερο όραμα ή στρατηγική. Αυτή ήταν η ΚΕΠΑ πάντα. Αυτό ήταν το βασικό μας κεφάλαιο εκκίνησης. Και εδώ έχουμε ανάμεικτα ε, αισθήματα. Ο πρόεδρος Μπρόκ ήταν πριν από τις ε, διαπραγματεύσεις. Η συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997 οδήγησε σε κοινέ στρατηγικές έτσι ώστε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο γεωγραφικό παράγοντα και να αποφασίσουμε για κοινέ δράσεις που θα απέρεαν από αυτήν. Και αφού ετέθησε εφαρμογή ε, η συνθήκη του Άμστερνταμ, τότε ε, επεκτείναμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, Ουκρανία και τη Μεσόγειο. Και ε, Πρόκειται για μια άμεσα αντίδραση σε μια συνθήκη η οποία εγκρίθηκε με βάση ε, κοινέ στρατηγικές. Μετά, ο ύπατος εκπρόσωπος, ο Χαβιέ Σολάνα, αξιολόγησε πολύ επικριτικά αυτές τις στρατηγικές, λέγοντας ότι δεν ε, ε, προέβαλαν προστιθέμενη αξία ε, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της ε, Βαρκελόνης και των διαφόρων συνθήκων και συμφωνιών. Επίσης είπε ότι επρόκειτο για καθαρά δηλωτικά κείμενα τα οποία δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητήθηκαν μέσω μιας διαδικασίας που αφορούσε μία προσέγγιση χριστουγεννιάτικου δέντρου, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να θέσουμε προτεραιότητες και να τις ιεραρχήσουμε. Και βασιστήκαμε σε βασικά διλήμματα και πολλές φορές μπορούσαμε να έχουμε σημεία τριβής με τους εξωτερικούς εταίρους. Γι' αυτό θέλαμε να ορίσουμε διαφορετικές προτεραιότητες και η στρατηγική του 2003 ήταν διαφορετική. Ε, επρόκειτο για ένα νέο έδαφος, για μια νέα προοπτική και δεν είχαμε ακολουθήσει τη διαδικασία επιτροπολογίες, επρόκειτο για ένα συγκεντρωτικό σχήμα τύπου κορεπέρ. Και ορίσαμε στόχους προτεραιότητες, ακόμα και ε, λανθάνουσες διαφορές με τους εταίρους, ξεκινώντας από τις ΙΠΑ. Αλλά ήταν ένα βασικό επίτευγμα μέσα από έκτακτες συνθήκες. Ο Σολάνα ήταν πολύ επιφυλακτικός να ακολουθήσει σχέδια δράσης για να μεταφέρει αυτή τη στρατηγική σε έμπρακτη δράση. Και όταν φτάσαμε σε μία πρώτη αναθεώρηση της στρατηγικής ασφαλείας το 2007, το 2008, είδαμε ότι ορισμένα ελληματικά στοιχεία, ορισμένα λατώματα ευρίσκονταν πάντα εκεί. Επρόκειτο για τις απειλές που θα μπορούσαν να πλήξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούσαμε να διαρθρώσουμε σωστά αυτές τις δυσκολίες και τις απειλές. Αυτή η διαδικασία εφαρμόστηκε και στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης που έχουμε με 10 εταίρους παγκοσμίω και πολλές φορές είναι δύσκολο να διαρθρώσουμε αυτές τις προτεραιότητες. Και στη συνθήκη της Λισαβόνας γίνεται λόγος για στρατηγικές στο άρθρο 26, όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αναγνωρίσει τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα οι ευέλικτες στρατηγικές ήταν οι πιο επιτυχείς. Η καταγραφή και συγγραφή των στρατηγικών είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και είναι πολύ δύσκολο να τις οριοθετήσουμε. Είτε θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα status quo που ήταν ένας μεγάλος κίνδυνος ή ίσως μπορούν να επέλθουν ε, ριζοσπαστικές αλλαγές όπως όρισε η κυβέρνηση Μπούς το 2002. Ήταν ε, μια πρόκληση σε σχέση με μια προγενέστερη συμπεριφορά τον είπα. Αυτό το μονοπάτι δεν είναι εύκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εμείς αποτελούμε ένα συνενετικό σχήμα. Το να σκεφτόμαστε στρατηγικά είναι ύψης της σημασίας. Και αυτό που έχει σημασία είναι να ελέγχουμε τις στάσεις και τα μονοπάτια που διανοίγονται. Ε, ζούμε σε ένα ε, κόσμο που μετασχηματίζεται με τάχιστους ρυθμούς μετά το 2003. Είναι, δεν είναι τόσο ευανάγνωστος αυτός ο κόσμος, ακόμα και στις γείτονες χώρες. Δηλαδή μιλάμε για το Μαλί, για το Αφγανιστάν, πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα χώρων, γειτονικών και μη που μας απασχολούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο ένα και χαμηλότερους συρρυκνούμενους πόρους εξαιτίας των περικοπών του προϋπολογισμού, της κρίσης της Ευρωζώνης, της χρηματοπιστωτικής κρίσης γενικότερα, καθώς και ε, των πολιτικών πόρων που όλο ένα και συρρυκνούνται βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλος διχασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υπάρχουν μεγαλύτερες προκλήσεις από το ε, εξωτερικό, δηλαδή υπάρχουν όλο ένα και διονγκούμενοι κίνδυνοι και αστάθεια, γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτά συμπεράσματα. Είναι δύσκολο να έχουμε μία σταθερή συνομιλία με εταίρους. Ο Καρλ Μπίλτ είπε ότι η όλη διαδικασία είναι πολύ πιο σημαντική από το τελικό προϊόν. Και γι' αυτό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς θα ορίσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη με βάση ε, ένα, μια σαφέστατη διαπραγματευτική εντολή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μισηρόλη. Πολλοί ζήτησαν το λόγο. Ο κύριος Κλίτς έχει το λόγο. Δεν ξέρω υπό ποια του ιδιότητα θα του δώσω το λόγο. Ο κύριος Κλίτς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τρέχουσα, τα τρέχοντα στρατηγικά συμφραζόμενα ε, αφορούν μία γενικότερη σύλληψη της στρατηγικής μας και η ασφάλεια διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία επινόησης μιας ε, στρατηγικής. Μέσα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ υπάρχει μια ε, στρατηγική στον τομέα της ασφάλειας, μέσα στα πλαίσια ε, μιας παγκόσμιας ασφάλειας και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που προείπαν οι κύριοι Μπίλτ και Σικόρσκι ο μεγαλύτερος ρόλος των νέων αναδυόμενων δυνάμεων, δηλαδή της ε, Κίνας και της Ρωσίας, που διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο. Έπειτα έχουμε αυτή τη δυναμική που διαγράφεται στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή Νομίζω ότι η Αραβική Επανάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαδικασία εκδημοκρατισμού και σταθερότητας σε αυτή την έφλεκτη περιοχή. Αλλά δυστυχώς επικρατεί το χειρότερο ε, σενάριο. Δυστυχώς οι φανατικοί Ισλαμιστές έχουν επικρατήσει και σε αυτές τις χώρες και στον δυτικό κόσμο. Ως προς τις σχέσεις με τις χώρες προς Ανατολάς, την γειτονία προς Ανατολάς βλέπουμε ότι η δημοκρατία και η σταθερότητα δεν είναι εξασφαλισμένη. Ως προς την πολιτική ασφαλεία στον ΙΠΑ βλέπουμε ότι από την Ευρώπη έχει μετατεθεί στον Ειρηνικό και στην Ασία. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την ΚΕΠΑ αλλά ίσως χρειάζεται ένα νέο έγγραφο περί στρατηγικής και μια ε, γενικότερη πολιτική ασφάλειας. Θα ήθελα να αναφέρω μερικούς παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Καταρχήν η Ευρώπη θα πρέπει να παρέχει από κοινού ασφάλεια. Θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και που κατέχουμε δυνάμει της συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης, καλύτερη, περισσότερη σταθερότητα και εκδημοκρατισμό στα Δυτικά Βαλκάνια μέσα στα πλαίσια της ενσωμάτωσής του στο ΝΑΤΟ. Επίσης, μεγαλύτερη ολοκλήρωση του κεφαλαίου της ασφάλειας και εκτενή ε, συνεισφορά μας στη Βόρεια Αφρική μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης στον τομέα της ασφάλειας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε εταιρική σχέση ασφάλειας με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ε, παρακολουθούμε την κατάσταση στη Γεωργία, στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρεμβαίνοντες για την εξαιρετική τους ε, εισήγηση και για την εργασία τους για την έγκριση αυτή της, ε, αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Θα πρέπει να είμαστε οξυδερκείς, όπως είπε και ο Υπουργός Σικόρσκι. Και νομίζω ότι ζούμε τη μεγαλύτερη κρίση μέχρι τούδε κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προφητείες, οι προφητείες όμως της απεσιοδοξίας δεν έχουν πληρωθεί. Η Ελλάδα δεν εγκατέλειψε την Ευρωζώνη, η Ιρλανδία έχει ανακάμψει μέσα στα πλαίσια της ε, Προεδρίας της και όπως είπε και ο Υπουργός Σικόρσκι ζούμε ε, σε μια κατάσταση ειρήνης ε, και σταθερότητας. Φτάσαμε σε μια μεγάλη αγορά 500 εκατομμυρίων, εκ των οποίων τα 300 εκατομμύρια χρησιμοποιούν το κοινό μας νόμισμα και είμαστε οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς και ε, πάροχοι υπηρεσιών. όλοι οι αναλυτές λένε ότι υπάρχει μια μετατόπιση του κέντρου βάρους προς ε, την Ινδία και τον Ειρηνικό. Θα ήθελα να σας πω ότι όλες οι μελέτες έλεγαν ότι η Ιαπωνία θα ξεπεράσει τις ΙΠΑ μέσα στα πλαίσια του ΑΕΠ. Είδαμε όμως ποια ήταν τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Μπίλτ μίλησε για, τις, ε, ε, για τη συνεισφορά των δεξαμενών ε, σκέψης. Αυτό μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε τους παράγοντες επιρροής. Οι ΙΠΑ λοιπόν επηρεάζουν επί τρία τον κόσμο σε σχέση με την Γαλλία, ε, Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα, καθώς και την Κίνα και την Ιαπωνία. Γιατί μιλάμε και για μικρά και για μεσαία κράτη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε και για τις ε, χώρες BRIC. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ε, μεγάλο μεταναστευτικό ε, κύμα. Η Δανία έχει ένα μεγάλο εξαγωγικό εμπόριο. Το ίδιο ισχύει για την Ινδία, το Λουξεμβούργο. Υποστηρίζει περισσότερο τα Ηνωμένα Έθνη από άλλες χώρες και η Ελλάδα ε, διαπρέπει στο εξωτερικό. Εάν όλα αυτά τα στοιχεία τα προβάλλουμε προς τα έξω βλέπουμε τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι αμεληταία η επιρροή μας. Όμως θα πρέπει να μπορέσουμε να επηρεάσουμε και τα παγκόσμια τεκτενόμενα ως προς το εξαγωγικό μας εμπόριο. Χτες, υπό την προεδρία του κυρίου Ντανζάν, μιλήσαμε για τις ανεπάρκειες της δράσης μας στον τομέα της ΚΕΠΑ, ότι υπάρχουν ελλείψεις δημοσιονομικού χαρακτήρα. Εμείς όμως έχουμε στείλει 1.800.000 στρατιώτες, δηλαδή 500.000 περισσότερους από τις ΗΠΑ και μπορούμε να αντλήσουμε πολλά διδάγματα από, την κρίση, από τις κρίσεις παγκοσμίως μεταξύ των οποίων και στη Λιβύη. Θα ήθελα να υποβάλω ε, ορισμένες, ε, ένα ερώτημα μάλλον προς τους Υπουργούς Εξωτερικών. Αυτή τη στιγμή αποτιμούμε τη δραστηριότητα της ΕΙΕΔ υπό τους Μπροκ και Γκουαλτιέρη. Θα ήθελα να ρωτήσω Ποιες αλλαγές ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να επέλθουν έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ε, μην προσυπογράφει τις μεγάλες κρίσεις, αλλά να μπορέσει να δράσει. Δηλαδή, όταν κάθεται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, όπως το Μέσα Ανατολικού, να μπορέσει να προβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές γειτονίες. Τι μας λείπει. Δεν υπάρχει πολιτική θέληση, υπάρχει επαρκώς πολιτική θέληση για να αντιμετωπίσουμε και τα δημοσιονομικά μας προβλήματα. Η εξωτερική μας πολιτική έχει γνωρίσει μία αύξηση του 3%. Τι μας λείπει όμως για να έχουμε ε, ενιαία φωνή στο παγκόσμιο στερέωμα, στη... στα Ηνωμένα Έθνη και ούτω καθεξής. πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με βάση τους μηχανισμούς που διαθέτουμε δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας, έτσι ώστε να ε, μετρήσει περισσότερο το ειδικό μας βάρος διεθνώς. Και οι δύο Υπουργοί έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες, έχουν πείρα και μπορούν να προωθήσουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εξωτερική μας πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος ε, Ράντεξ Σικόρσκι μίλησε για κάποια στατιστικά από το παγκόσμιο εμπόριο. Εγώ ήθελα να αναφερθώ και στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Τελευταία, οι ΙΠΑ κάλυπταν το 50% όλου του, όλων των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ και τώρα καλύπτει το 25%. Ως Ευρωπαίοι, και αναφέρθηκε εδώ, αλλά νομίζω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να σοβαρευτούμε. Δηλαδή, θα δούμε μόνο την ήπια δύναμή μας στον κόσμο ή ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουμε παρουσία παντού. Διότι λόγω των προβλημάτων των Αμερικανών θα μειωθεί η συμβολή τους στις αμυντικές δαπάνες. Αυτό θα το δεχτούμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Θα πούμε εντάξει συνεχίζουμε ως έχουμε ή θα πούμε ότι χρειάζεται όχι μόνο ήπια δύναμη αλλά και άσκηση ισχύω με πιο ε, επιθετικά μέσα όπως στη Λιβύη ή αλλού ή όταν θέλουμε να φροντίσουμε ε, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η σταθερότητα ή να βρεθεί πολιτική συμφωνία στη Βοσνία Ερζεγοβίνη ούτως ώστε να μπορέσει η διεύρυνση να συμπεριλάβει στη βοσνια ζεγοβινη ουτως ωστε να μπορεσει η διευρυνση να συμπεριλαβει ολα τα Δυτικά Βαλκάνια. Και υπάρχει και το θέμα των ε, αβεβαιοτήτων στα σύνορα. Μιλήσαμε για την ε, ανατολική γειτονική διάσταση. Εκεί υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν μεγάλες δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ τους. Και εμείς ως Ευρωπαίοι κάποια στιγμή μπορεί να κληθούμε να έχουμε δυνάμεις ε, σταθεροποίησης ή παρακολούθησης σε αυτές τις δύσκολες περιοχές. Μπορούμε να το κάνουμε ή είμαστε διατεθειμένοι να ε, διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των δικών μας ανθρώπων προκειμένου να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της σταθερότητας σε κάποιες περιοχές. Έγιναν αναφορές και στις αλλαγές στη Βόρεια Αφρική και την Αραβική Άνοιξη, τον Αραβικό χειμώνα ή τέλος πάντων τι είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα. Καμιά φορά είμαστε υπεραισιόδοξοι Χρειάστηκαν δεκαετίες για να μην πω αιώνες ώστε η Ευρώπη να φτάσει στη θέση που είναι σήμερα. Δηλαδή γιατί πρέπει να περιμένουμε ότι ε, χώρες που δεν γνώρισαν ποτέ τη δημοκρατία θα μπορέσουν σε ένα συντομότατο χρονικό διάστημα να περάσουν μέσα από αυτό τον καταπληκτικό μετασχηματισμό που έλαβε χώρα στην ε, Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη σε δεκαετίες. Γιατί χώρες όπως η Αίγυπτος ή άλλες βορειοαφρικανικές χώρες ε, θα ακολουθήσουν ε, αλλαγές πολύ γρήγορα όπως οι ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες που όμως είχαν ένα ε, συγκεκριμένο όραμα και συγκεκριμένο προσανατολισμό, είχαν στόχευση που δεν έχουν οι χώρες της Βόρειας Αφρικής. Μας περιμένει μια δύσκολη περίοδος. Τι θα κάνουμε συγκεκριμένα. Και ξαναγυρίζω στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Με αυτό άρχισα. Έχουμε πρόβλημα γιατί έχουμε την Τουρκία, την Κύπρο και άλλα προβλήματα που πρέπει επίσης να μπορέσουμε να τα λύσουμε αν θέλουμε αποτελεσματική άμυνα και αποτελεσματική ασφάλεια. Thank you. Mr. Κυρία Γκόμες, κυρία Μπίλτ. Συρία είναι αποτυχία της Ευρώπης και του κόσμου να λάβει την ευθύνη να προστατεύσει τους ανθρώπους και κάποιους κανόνες να τους εφαρμόσει. Μπορούμε να είμαστε εμείς παγκοσμίω ένας αξιόπιστος φορέας για την ειρήνη, εάν δεν θέσουμε το θέμα της νομιμότητας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και εάν δεν έχουμε μία θέση μονίμου αντιπροσώπου του Συμβουλίου Ασφαλείας και δεν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Γιατί τώρα η Σουηδία είναι αντίθετη προς ε, προσφυγή στο ε, δικαστήριο σε όλους ενέχονται σε εγκλήματα στην Συρία. Αναφέρατε δεν τις πυρώσεις, τα Όλα αυτά υπάρχουν στη συνθήκη της Λισαβόνας. Η ύπατη εκπρόσωπος είναι αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έπρεπε να ότι η Επιτροπή και διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται με τα θέματα της ενέργειας του εμπορίου κάνουν κάτι και στα πλαίσια εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι θέμα μόνο συμφερόντων, είναι θέμα απειλής και της δικής μας ασφαλείας. Δεν είναι λοιπόν εκπληκτικό το ότι οι υπουργοί μας δεν μπορούν να συμφωνήσουν ακόμη και σε θέματα κοινή ε, χρηματοδότησης των αποστολών που στέλνουμε στην περιοχή του Σαχέλ και ε, στο Μαλί. Στο Μαλί. Σε μια τέτοιου είδους μη στρατιωτική αποστολή. Δεν είναι εκπληκτικό το ότι έτσι όπως πήρε αποφάσει το Συμβούλιο δεν ε, έχει καμία φιλοδοξία ακόμη και για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μήπως δίνει λάθος μηνύματα, όχι μόνο στους πολίτες μας αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Κύριε Μισηρόλη, δεν είναι μόνο θέμα ταυτοποίηση των στρατηγικών συμφερόντων. Και στρατηγική υπάρχει, αλλά μήπως χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική ηγεσία Μήπως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των πολιτών της Ευρώπης και όχι για ολίγων. Δεν πρέπει να αρχίσουμε να νοικοκυρεύουμε ε, εμείς πρώτα απ' όλα την Ευρώπη μας πριν να δούμε τι θα κάνουμε για τον υπόλοιπο κόσμο. the floor has, uh, Mr. Κύριε Σέμπιτ, αν το προφέρω καλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου άρεσε η μεταφορά του κυρίου Σικόρσκι για το hardware και το software, αλλά όταν μιλάμε για την αποτελεσματικότητα του software, πρέπει να σκεφτούμε και την ανάπτυξη του hardware. Τι θα γίνει το hardware. Πώς πεθαίνει ένας ε, πολιτισμός είναι ένα βιβλίο που θα ήθελα να παραθέσω στο τέλος του αιώνα ε, θεωρώντας ότι θα υπάρχει ε, συνεχής ανάπτυξη ο πληθυσμός της Δυτικής Ευρώπης από ηλικία 50 μέχρι 59 ετών θα μειωθεί κατά 2,5 και κατά 2 τρίτα στην Ανατολική Ασία ο πληθυσμός, ο ενεργός πληθυσμός στον ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά ένα τέταρτο. Οι λιγότερο γόνιμες ευρωπαϊκές χώρες, οι πιο βιομηχανικές βέβαια, θα δουν να μειώνεται ο πληθυσμός του συνολικά 40 με 60% ε, κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα. Αυτή είναι μια ιστορία που δεν ε, προβάλλεται είναι το δημογραφικό πρόβλημα σε όλο το βιομηχανικό κόσμο που απειλεί να στρεβλώσει την ε, παγκόσμια οικονομία και τη σταθερότητα. Η Ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ρωσία ήδη αντιμετωπίζουν ε, ένα τεράστιο πρόβλημα στην εξέλιξη ε, του δημογραφικού. Όταν μιλάμε κυρίες και κύριοι για στρατηγική του μέλλοντος και αυτό θέλω να πω, εκεί θέλω να καταλήξω, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα δημογραφικά στοιχεία και τις εξελίξεις. Αλλιώς πρόκειται να απογοητευθούμε πάρα πολύ. Δεν θα ε, λειτουργήσει το software γιατί δεν θα έχουμε hardware. Άλλη παρατήρηση τώρα. Δεν μου φαίνεται να έχει νόημα να βλέπουμε την Ευρώπη ως υπερδύναμη με στρατιωτικές δαπάνες που είναι στο 1% του ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες. Γιατί γι' αυτό ε, δημιουργήσαμε και τον όρο soft power, πια δύναμη, για να καλύψουμε το γεγονός ότι από στρατιωτικής άποψης είναι αδύναμη η Ευρώπη. Soft power δεν υπάρχει. Και αν η Ευρώπη δεν μπορέσει να έχει πραγματική δύναμη να ε, προβάλλει την ισχύ της εκτός των συνόρων της Ευρώπης, δεν θα είναι ε, ε, δύναμη μεγάλη. Ίσως οικονομικά να είναι, αλλά στρατιωτικά όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω συμμερίζομαι αυτά τα οποία λέξαν για τις φιλοδοξίες μας, αλλά χωρίς να Θέλω να κάνω παρατηρήσεις ε, πάρα πολύ απλές. Όπως είπε και η Άννα Γκόμες, πολλά πράγματα υπάρχουν ήδη στη συνθήκη της Εσόνες. Πολλά υπάρχουν ήδη στις συμφωνίες που έχουν ε, γίνει ε, σε επίπεδο συμφωνιών συμβουλίου, όπως τα headline goals Έχουμε πάρα πολλά μέσα και εργασία, μηχανισμούς, φιλοδοξίες, θεσμικά όργανα, πολλά στη διάθεσή μας, ήδη. Λείπει συνεκτική και συνενετική πολιτική βούληση για να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Και επιτρέψτε μου να πω το εξής. Με μεγάλη μου έκπληξη πάντα διαπιστώνω ότι κάθε έξι μήνες γίνονται, γίνεται μία άτυπη συνάντηση για θέματα άμυνας. Λιγότερο από 1 τρίτο των υπουργών παρίσταται. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Μαλί τι γίνεται. Ένα κρατός μέλος υποστηρίζει τη χώρα αυτή. Όλοι λένε ότι υποστηρίζουν αυτή τη χώρα αλλά λιγότερο από τους μισούς εκπροσωπούνται στο επίπεδο που πρέπει να συζητηθούν κάποια πράγματα, στο επίπεδο της πούληση της πολιτικής. Γιατί εκεί πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Ξέρουμε βεβαίως καλύτερα από όλους ότι είναι πάρα πολύ φορτωμένη η ατζέντα των υποχρεώσεων όλων. Και πολλές φορές βλέπω οι πολίτε, ευτυχώ που δεν βλέπουν τον κατάλογο παρόντων στι συνεδριάσει στα διάφορα θεσμικά όργανα που πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις και οι πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον, την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Τώρα, αυτό το είπα εν παρενθέσει, αλλά σοβαρά θα πρέπει να πω. Δεν χρειάζεται κάθε έξι μήνες να ανακαλύπτουμε την πυρά και να αρχίζουμε με ωραίες συζητήσεις. Έχουμε τα κατάλληλα μέσα, πρέπει όμως πολιτική βούληση για να τα θέσουμε σε εφαρμογή ο καθένας πρέπει να επομιστεί τις ευθύνε τους οι πάντες και οι υπουργοί σε κάθε χώρα μέλος για να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο γερουσιαστής κύριος Κλής. Οι στατιστικές του κυρίου Σαλαμφράγκα είναι πολύ χρήσιμες. Πολλά μέλη ανέφεραν το θέμα των δυνατοτήτων που έχουμε στον τομέα της άμυνας, κυρίως σε σύγκριση με αυτές που διαθέτει, διαθέτουν οι ΙΠΑ. Ε, σε επίπεδο δαπανών αμυντικών δαπανούμε σχεδόν το 1 τρίτο σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και νομίζω ότι εάν είχαμε για τα χρήματα αυτά που δαπανούμε και το 1 τρίτο των δυνατοτήτων, καλά θα ήταν. Αν δείτε όμως τα αποτελέσματα είναι χειρότερα. Κάποιος ανέφερε ότι έχουμε ένα κόμμα, ε, ένα εκατομμύριο ε, χιλιάδες ε, στρατιώτες αν την Ευρώπη. Αναπτύσσουμε μόνο το 6% αυτό που διαθέτουμε. Φανταστείτε αν είχαν οι ΙΠΑ, αν είχαν 50 επιτελεία, 50 διαφορετικές, ε, διαφορετικά επιτελεία για το, τον στρατό ξηρά θαλάσσης για την αεροπορία και 50 διαφορετικά συστήματα. Η πρότασή μου λοιπόν θα είναι, όταν αρχίζουμε νέα προγράμματα, φερρυπίν, για τις μη επανδρομένες δυνατότητες, να δούμε και τις δημόσιες συμβάσεις. Όταν έχουμε χιλιάδες επιχειρήσεις που κάνουν τα ίδια πράγματα, κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε και ομαδοποιήσεις αυτών των δημοσίων αγορών, ώστε να κάνουμε καλύτερα για τον καθένα μας ε, τη δουλειά μας και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά αυτά όλα απαιτούν πολιτική βούληση, που δεν υπάρχει πάντα. Στα λόγια είμαστε καλοί. Λέμε ότι θέλουμε να ενεργήσουμε από κοινού, αλλά στην ώρα της πρακτικής εφαρμογής βεβαίως υπερισχύουν τα εθνικά συμφέροντα πάνω απ' όλα. Και για θέματα όπως εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανώσεις, τι ανέφερε κυρία Γκόμες, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πράγμα το οποίο με κάνει στο να πω ότι βλέπουμε εδώ την απεικόνηση αυτής ε, των γεγονότων εδώ. Η Πολωνία υποστήριξε την υποψηφιότητα της Γερμανίας. Ο Έλμαρ όμως μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Πράγμα το οποίο πραγματικά μας δίνει μια σαφή εικόνα του προβλήματος που υπάρχει. Υπάρχουν στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών πολλές θέσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο αποδοτικοί εάν εκπροσωπούμεθα από κοινού. Και το ερώτημα είναι, είμαστε πιο ισχυροί αν σε επίπεδο ΠΟΕ μας εκπροσωπεί μόνο η Κομισιόν και όχι τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι κάτι πως λογική μπορεί να ισχύσει και για άλλες διεθνείς οργανώσεις. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε δισεκατομμύρια εάν ως κράτη-μέλη δεν εκπροσωπούμεθα πλέον στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι, όπως σήμερα, αλλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η αλήθεια ποια είναι. Θέλουμε να ενεργήσουμε από κοινού, με μία φωνή. Ή να το συζητάμε. Αν δεν κάνουμε κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι. I agree with Mr. Gapes that, um... Συμφωνώ με τον κύριο Γκέιπς ότι Ίσως δεν έχει γίνει η δουλειά που έπρεπε να έχει γίνει στα Βαλκάνια, έπρεπε να έχουμε παρέμβει ίσως αλλού και ίσως στον περιοχή του Καυκάσου και ίσως επαναλάβουμε τις αποτυχίες μας και στον στρατιωτικό τομέα με καταστροφικό τρόπο, όπως το κάνουμε και στο νομισματικό. Ξέρουμε ότι δεν ήταν θετικό το σύμφωνο σταθερότητος. Στην ώρα της αλήθειας, έξι φορές είδαμε ότι είχαμε τους κατάλληλους μηχανισμούς για να επιτύχουμε, δεν είχαμε τις κατάλληλες ε, διαδικασίες και καταλήξαμε σε πολύ μεγάλες κρίσεις. Στο στρατιωτικό τομέα ίσως το χτύπημα να είναι πολύ πιο απότομο και πολύ πιο σοβαρό από ό,τι στον τομέα τον οικονομικό. Και υπάρχουν σημεία προειδοποίησης παντού. Ακόμη δεν έχουμε μάθει τα μαθήματα, τις αδυναμίες που επιδείξαμε στα Βαλκάνια τη δεκαετία των 90 και συμμερίζομαι την απογοήτευσή σας για την έλλειψη αρκετής συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Οι άνθρωποι μας πεθαίνουν διότι δύο οργανώσεις στις οποίες τα περισσότερα μέλη είναι κοινά, δεν μπορούν να αλληλοβοηθηθούν. Πριν από κάποια χρόνια, νόμιζα ότι είχα τη λογική ιδέα να συστήσω πέντε ο ευρωπαϊκές ομάδες ανασυγκρότησης σε κάποιες περιοχές του Αφγανιστάν, για να φέρω αυτό το παράδειγμα. Όταν το κλίμα ήταν πάρα πολύ θερμό στη νότια περιοχή. Χρησιμοποιώντας κάποιους πόρους αναπτυξιακούς θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τους ε, θανάτους αυτές τις πολύ καυτές περιοχές. Αυτό όμως απέβει αδύνατον διότι έπρεπε να υπάρχει η προστασία των, δυνα... δυνάμεων του ΝΑΤΟ και κάποια πράγματα δεν... τα μπορούσαν να γίνουν εξαιτία του προβλήματος που υπάρχει στην Κύπρο. Υπάρχουν ε, εκλογές τώρα. Δεύτερος κύκλος εκλογών στην Κύπρο την Κυριακή. Ελπίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα μπορέσει να αλλάξει κάποια πράγματα το status quo πραγματικά δεν είναι σωστό. κυρία Γκόμες είπε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κοινή χρηματοδότηση για το Μαλί. Τι ακριβώς εννοείται. Δεν θυμούμε καλά τους αριθμούς. Από ό,τι θυμούμε έχουμε προβλέψει τις αφρικανικές δυνάμεις 50 εκατομμύρια και σε θέματα αναπτυξιακής βοήθειας άλλα 200. Τι εννοείται. Χρηματοδότηση της ε, επιχείρησης ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να παραλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος και να μην αντιγράψουμε τα σφάλματα του ΝΑΤΟ που χρηματοδοτήθηκε για πόλεμο παντού. Τώρα όμως έχουμε άλλου είδους επιλογές. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε κίνητρα με τρόπο που να οδηγήσει αυτούς που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους αποστολές ε, να τα δίνουν όλα και άλλοι που δεν συμμετέχουν να εξοικονομούν χρήματα. Διαφορετικά θα πρέπει να τα πράγματα. Και ο κύριος Σέμπη σωστά τα ότι είπε για την ε, μείωση του πληθυσμού. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι σοβαρό και αυτό που είναι ενισχυτικό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ λίγα μέσα για να επηρεάσουμε την κατάσταση. Τα άτομα για τα οποία μιλάτε έχουν ήδη γεννηθεί. Υπάρχουν γενιές οι οποίες δεν βρίσκονται πλέον στην ε, παραγωγική ηλικία which are politically difficult. Um, υπάρχουν και εδώ δυσκολίες. Αλλά και αυτό είναι ένα επιχείρημα που θα πρέπει να μας κάνει να συσπηρωθούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε επίτηδες. Βεβαίως, όπως ελέγχθη, υπάρχουν τα μέσα στις συνθήκες για να ενεργήσουμε και το πραγματική δοκιμή θα είναι αν πραγματικά οι μεγάλες χώρες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα και τα εργαλεία που υπάρχουν για να υλοποιήσουν αυτά τα οποία προβλέπουν οι συνθήκες. leadership... Κυρία ε, Γκόμες, όταν μιλάμε για πολιτική ηγεσία, τότε οι αναλυτές δεν θα πρέπει να έχουν το λόγο, αλλά οι πολιτικοί. Γιατί υπάρχει και ένα στοιχείο ε, νομιμότητας και εντολής από τους πολίτες. Εάν κοιτάξουμε προς τα πίσω, Λίγα χρόνια πριν, οι πολίτες μας δεν μας είχαν ζητήσει να δράσουμε ε, κατά δραστικό τρόπο. Είχαμε το μάντρα της δεκαετίας του 90, το οποίο όμως δεν είχε εισακούστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικοί έπρεπε να το λάβουν υπόψη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έπρεπε να δράσει και να αποφασίσει ως προς τη στρατηγική μας δράση. Και αν δούμε την ατζέντα μας των τελευταίων 15-20 συνεδριάσεων, βλέπουμε ότι η ΚΕΠΑ ήταν υψηλά στην ε, ατζέντα. η πολιτική μας όμως είχαν και άλλες υποχρεώσεις. Στο τέλος του μήνα προβλέπεται μία συνάντηση, αλλά Ίσως η συνθήκη της ε, ε, Λισαβόνας οδήγησε στο να μην ε, προσκαλούνται πάντα Υπουργοί Εξωτερικών για συζητήσεις τέτοιας υφής. Υπάρχουν πολλές προσδοκίες από το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας αργότερα κατά το τρέχον έτος. Το στοιχείο της άμυνας ανέκυψε διότι θα πρέπει να αποφασίσουμε για το τι θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλους εταίρους, το ΝΑΤΟ, ΙΠΑ και την Αφρικανική Ένωση. Αυτός είναι ένας φυσικός εταίρος στην περίπτωση του Μάλι αλλά τα στρατιωτικά και αμυντικά ζητήματα δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε απομονωμένα. Θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση γιατί έχουμε και άλλα μέσα στη διάθεσή μας και εδώ έγκυται η προστιθέμενη αξία. Δηλαδή πέρα από τα θεσμικά όργανα και την πολιτική θέληση θα πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι. Και όταν υπάρχει πολιτική θέληση και τα άρθρα της συνθήκης να είμαστε ετοιμοπόλεμη, να το πω έτσι. Και αυτό αφορά και το λογισμικό και τον εξοπλισμό μας, το hardware. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Πόλετς. Α, όχι. Θα απαντήσει ο κύριος Μπίλτ. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί συμφωνώ με όλα όσα ακούσαμε. Κάποιοι προβληματισμοί μόνο επί ορισμένων θεμάτων. Τώρα, για το θέμα των μέσων και δυνατοτήτων στην άμυνα, συμφωνώ με αυτά που είπατε, αλλά να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι μια μεγάλη μετατόπιση στον ε, τρόπο με τον οποίο ε, σχεδιάζουμε τις δυνάμεις μας. Πάμε, πήγαμε σε πολλές χώρες ε, όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε μεγάλες αμυντικές δομές στο παρελθόν, τώρα έχουμε δομές πιο εξαρτευτικές, εξαρτευτικού σώματος. Πριν από πολύ καιρό αρχίσαμε τη δεκαετία του 50 ε, και έχουμε και στρατό σε περιφέρειες, αλλά τώρα είναι εξτρατευτικά σώματα. Πριν από 15 χρόνια και οι Γάλλοι είχαν παρόμοια εμπειρία ε, η δομή τους όμως μειώθηκε γιατί δεν ε, χρειάστηκε. Και στη Σουηδία συνέβη το ίδιο. Παλιά είχαμε πολύ περισσότερο στρατό, τώρα έχουμε μικρότερες, λιγότερες δυνάμεις, αλλά με περισσότερες ε, δυνατότητες. Οπότε αριθμητικά βλέπουμε να μειώνονται οι, οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά είναι περισσότερες οι εκστρατευτικές δυνατότητες. Ε, αρκεί αυτό όταν υπάρχει κάποια ένοπλη σύγκρουση. Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα σημειώθηκε αυτή η αλλαγή. Αυτό δεν το βλέπουν οι Αμερικανοί, γιατί δεν πέρασαν ε, από τέτοιες εμπειρίες. Ε, δεν υπήρχαν δηλαδή περιφερειακοί πόλεμοι, μόνο κάποιες συγκρούσεις ε, στα σύνορα Μεξικού-Τέξας. Ε, ενώ στην Ευρώπη υπήρχαν περιφερειακοί ε, πόλεμοι εδώ και χρόνια. Σε ό,τι αφορά τα μέσα και δυνατότητές μας, σίγουρα χρειαζόμαστε και πιο σκληρή δύναμη. Αναφέρθηκε η Λιβύη. Νομίζω το έχω ξαναπεί και εδώ μπροστά σας. Με απασχολεί περισσότερο η έλλειψή μας στη διπλωματία παρά στην άμυνα. Η Λιβύη, η Λιβύη ως παράδειγμα. έχουμε τη δυνατότητα να ρίξουμε το καθεστώς. Μπορούμε να ε, ρίξουμε καθεστώτα αν θέλουμε και με την βοήθεια των Αμερικανών για να μην ε, ε, έχουμε επικαλύψεις δυνάμεων. Μπορεί να γίνει αυτό, είναι εφικτό. Το δύσκολο όμως δεν είναι να ρίξουμε αλλά να οικοδομήσουμε καθεστώτα. Κοιτάξτε τη Λιβύη σήμερα. Από τη Βενγάζη έπρεπε να τους κενώσουμε όλους. Δεν έχουμε πρόσβαση πια εκεί. Ε, βλέπουμε να εξαφανίζονται τα σύνορα, βλέπουμε όπλα παντού, ε, βλέπουμε aftershock ε, στο Μαλί και σε άλλες χώρες και που ξέρουμε, δεν ξέρουμε πού αλλού. μπορεί να γίνει κάποια παρακολούθηση των συνόρων ή να υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις, αλλά υπάρχει δυνατότητα σε επίπεδο διπλωματικό και αναπτυξιακό, ούτω ώστε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου δημοκρατικού κράτους στη Λιβύη εύκολα καταστρέφεις. Μπορείς όμως να ε, οικοδομείς, να ανοικοδομείς. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε επιτυχία στο Αφγανιστάν. Ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση εδώ. Δεν καταφέραμε να επανενώσουμε μετά από τόσα χρόνια την Κύπρο. Ε, αυτή είναι μια διπλωματική έλλειψη εκεί, παρόλο που είχαμε δυνατότητα ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπερδινιστερία κάναμε ε, μια ε, αποστολή πολιτισμική μάλλον θα λέγαμε, πολιτιστική. Ξέρετε πού είναι, έχετε πάει. Είναι ένας θύλακας στην Ευρώπη που έχει μείνει από τη Σοβιετική περίοδο όπου περνάμε από ε, ε βλέποντας σημαίες με σφυροδρέπανα και μπαίνουμε σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Δεν έχετε πάει. Πρέπει λοιπόν να αφιερώσουμε μέσα διπλωματίας και μέσα για την επίλυση διαφορών σε πολλούς τομείς. Ακόμα ε, οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Έχουμε προκλήσεις ε, στα Βαλκάνια και αλλού. Ε, τι γίνεται όμως στην Ανατολή. βλέπουμε ότι ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται συνεχώς. Πάμε δηλαδή ε, μέχρι, πάμε για μια μεγάλη καταστροφή ε, από το ε, Λίβανο μέχρι την Μπάσρα. Έχουμε τις δυνατότητες, τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε την καταστροφή. Μπορούμε να συζητούμε αενάως για ε, κυρώσεις, ICC κλπ. Εδώ όμως θα πρέπει να ε, συγκληθεί Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να αναλάβει δράση, να σταματήσει ε, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες για να υπάρξει μια πρώτη σταθεροποίηση, πράγμα πολύ δύσκολο, και βεβαίως ε, και το θέμα του ICC, δηλαδή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της δικαιοσύνης. Ε, να έχουμε πρόβλημα 16 χρόνια μετά τον πόλεμο της Βοσνίας. Τώρα η προτεραιότητα πια είναι να τελειώσει ο πόλεμος, να τελειώσουν οι σφαγές και μετά θα προχωρήσουμε στο επόμενο ε, στάδιο. Εάν πάμε να τα κάνουμε όλα μαζί, είμαστε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις που μας περιμένουν ή κάποιες μεγάλες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Έχουμε τα μέσα, τους μηχανισμούς για τη σταθερότητα, για την επιβολή του κράτους δικαίου, για την ανασυγκρότηση κρατών, ε, χωρών μετά από τεράστιες ένοπλες συγκρούσεις και καταστροφές κοινωνιών. Και δεν μιλάω εδώ για καταστροφή κτηρίων. Ούτε τόσο, αν θέλετε, δεν, δεν αναφέρομαι τόσο στα θύματα εδώ, όσο στο, στον κοινωνικό ιστό που καταστρέφεται. Γιατί ε, η σύγκρουση, αυτή η σφοδρή σύγκρουση κρατών ε, δημιουργεί καταστροφές που παίρνουν χρόνο για να ε, αποκατασταθούν. Ε, ε, κράτη-μέλη της Ένωσης έχουμε ε, συμμετάσχει σε διπλωματικό επίπεδο με κάμια 60 χιλιάδες. Αν υπολογίσουμε τις ανθρωποώρες που αφιερώνουν οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες σε ίσονο σημασία εκδηλώσεις, αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σωστά και αν χρησιμοποιούνταν σωστά θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της Λιβύης. Ε, πολλές φορές ε, οι πόροι μας είναι βέβαια και περιορισμένοι. Γι' αυτό χρειάζονται σύντονες προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο. Γιατί ο καθένας μας από μόνος του ε, δεν ε, έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ε, Τώρα αρχίζουμε να αναπτύσσουμε νέα μέσα και μηχανισμούς. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό ε, Ίδρυμα Ινστιτούτο για την Ειρήνη, νέο. Χρειαζόμαστε μέσα προληπτικής δημοκρατίας, ε, διπλωματίας, γνήσιας διπλωματίας, ε, επίλυσης διαφορών. Βεβαίως ε, δεν είμαι κατά ε, αυτού που χρειάζεται για να βελτιώσουμε την αμυντική μας ικανότητα, αλλά με ενδιαφέρει πιο πολύ να κλείσουν τα κενά στο τομέα της διπλωματίας και στη δυνατότητα συμβολής στην ανασυγκρότηση, ιδιαίτερα ε, όταν σκέπτομαι ότι τις επόμενες δεκαετίες θα υπάρξουν πολλές αναταράξεις και συγκρούσεις στις ε, ε, γειτονικές μας περιφέρειες και ε, βλέποντας βέβαια και τα ανεπίλητα προβλήματα, βλέπω Κυπριακό, Αφγανιστάν, αλλά και τώρα τα καινούρια Συρία, Μαλή, και η πραγματική πρόκληση μπορεί να είναι αλλού. Δηλαδή, ο πραγματικός, η πραγματική απειλή ασφαλείας θα μπορούσε να προέλθει από αλλού. Ε, ας πούμε, από τον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ, κύριε Πόλιτ. Ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στους δύο υπουργούς για την ε, αυτή πολύ βασική εισαγωγή στην προβληματική μας και τη συζήτηση. Ε, είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμβάλλει στην ειρήνη και την ευημερία και μέσα από την ε, ενιαία αγορά, αλλά θα πρέπει να δώσουμε απάντηση και στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και του πολυπολικού κόσμου με τους Κινέζους, με τα δισεκατομμύρια τους, τους Ινδούς, με τα δισεκατομμύρια πληθυσμού, αλλά και τον Πόλο, των Ήπα. Χρειάζεται λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού να έχουμε κοινή δράση προς τα έξω. Και έτσι θα ε, προασπίσουμε και τα εθνικά μας αλλά και τα κοινά μας πάνω απ' όλα συμφέροντα. Γι' αυτό πρέπει να βλέπουμε με ενιαίο τρόπο τα πράγματα. Έχουμε δυνατότητα συντονισμού των απόψεων ε, μέσα από πολιτικές επιτροπές, από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, αλλά από ό,τι βλέπω και παρατηρώ, όλα αυτά κατά κανόνα οδηγούν σε μια πολιτική αντίδρασης και όχι πρόληψης και δράσης. Αν δούμε τι θέλουμε να επιτύχουμε στον κόσμο, δηλαδή ποια είναι, ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας, για να ε, τους επιτύχουμε χρειαζόμαστε στρατηγική. Πρέπει λοιπόν να συνενώσουμε τις ε, ικανότητες που έχουμε, τους διπλωμάτες, ε, αυτό που είπε ο κύριος Μπίλντε ε, δεν το ήξερα σχετικά με τον αριθμό των διπλωματών που ε, δραστηριοποιούνται και χρειάζεται και δικτύωση των ικανοτήτων μας. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική που εξετάζουμε τώρα είναι πολύ χρήσιμη, ήδη έχουν διατυπωθεί οι πρώτες ιδέες σχετικά, πρέπει όμως ε, να επεξεργαστούμε και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, γιατί από τότε που πρώτο διατυπώθηκε άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Συμφωνώ με τον Κάρλ Μπίλτ, ιδιαίτερα ε, με αυτό που είπε στην δεύτερη παρέμβασή του, ότι η εξωτερική πολιτική της Ένωσης είναι κάτι πολύ παραπάνω από στρατιωτικές επεμβάσεις. Όμως ε, η χρήση στρατιωτικών μέσων ως τελευταίο ίστατο μέσο καταφυγής ε, πρέπει να συγκαταλέγεται στις δυνατότητές μας. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα επηρεαστούν όλα αυτά από μια κοινή εξωτερική πολιτική, γιατί η χρήση στρατιωτικών μέσων βεβαίως εδώ άπτεται της κεντρικής μας αντίληψης περί κυριαρχίας. Και αναφέρθηκε ότι ε, χρειάζεται το pooling και sharing, δηλαδή η συνένωση και κοινή χρήση των δυνάμεων. Και αν τα δούμε όλα αυτά, πάμε στο αμέσως επόμενο ε, ερώτημα. Πώς μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κάτι από κοινού και ένα σημαντικό κράτος μέλος το οποίο ε, καλείται να διαθέσει ικανότητες μέσα και δυνατότητες που έχει και που διακρίνεται σε αυτά και δεν θέλει και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό δεν θα είναι η απαρχή της ε, αποτυχίας αυτής της κοινή προσέγγισης. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Και χθε στο Βερολίνο είχαμε μια ακρόαση ε, για ε, την ΚΕΠΑ όπου συζητήσαμε για την ε, συνένωση και την κοινή χρήση των πόρων. Βεβαίω υπό εθνικό έλεγχο η συμβολή της κάθε χώρας ελέγχεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις αποστολές και που λαμβάνουν χώρα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Όπως έδειξε και η περίπτωση του Μαλή, θα πρέπει να υπάρχει γρήγορη διαθεσιμότητα όλων αυτών των δυνάμεων. Δεν τα καταφέραμε τόσο πολύ στο Μαλή. Βέβαια, με την προετοιμασία της εκπαιδευτικής αποστολής ε, μπορέσαμε από κοινού να κρίνουμε την πολιτική κατάσταση, τις, τις ανάγκες της χώρας και εκεί κινηθήκαμε πιο γρήγορα στο Μαλή. Ε, βεβαίως ε, η Γαλλία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο εκεί. Τώρα, για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και την επανεξέταση της στρατηγικής αυτής, θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε μια διαδικασία όπως έκανε το ΝΑΤΟ, όπου η Μάντλεν Ολμπράιτε έκανε, δημιούργησε ομάδα εμπειρογνωμόνων για να κλείσει το κενό μεταξύ εμπειρογνωμόνων και διπλωματίας. Χρειαζόμαστε και εμείς μια τέτοια κοινή ε, συζήτηση για τη στρατηγική πάνω σε κοινέ βάσεις, ούτως ώστε να συγκεράσουμε και τις διαφορετικές μας ε, νοοτροπίες ε, και ε, απόψεις. Μια ανάπτυξη στρατηγικής δεν συνεπάγεται ένα νέο κείμενο, αλλά και μετά από 10 χρόνια ένα καινούργιο τρίτο ε, έγγραφο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ε, συνεχής διαδικασία. Σε ορισμένα δύσκολα θέματα πρέπει να πούμε από την άλλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλή στρατηγική ασφάλειας. Βλέπε η Ιράν, όπου και στο πυρηνικό θέμα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις δηλαδή για τα πυρηνικά της χώρας αυτής και έχει λόγο και για θέματα συνεργασίας και για θέματα επιβολής κυρώσεων στο Ιράν ενδεχομένως. Ελπίζω ότι όλα αυτά σύντομα θα στεφθούν από την ε, επιτυχία που περιμένουμε. Έχουμε πολλούς ομιλητές. Μπορούμε να περιοριστούμε στα δύο λεπτά. Έτσι μόνο θα μιλήσουν όλοι. Ο κύριος Βάιγκελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Στα δύο λεπτά θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Καρλ Μπίλτ για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ε, αναφέρθηκε στη Συρία μεταξύ άλλων με μεγάλη απογοήτευση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πόσο πια, πόσα μπορούμε να καταπιούμε, ποιο είναι το αντίτιμο της καταστροφής ενός κράτους και της απομάκρυνσης ενός καθεστώτος που δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να βρεθούμε σε κατάστασεις όπου το αντίτιμο να είναι τόσο υψηλό και στο, στη Συρία βρισκόμαστε σε αυτή ακριβώς την κατάσταση, πολύ κοντά σε αυτό. Αυτό που έχει σημασία, όπως και στο κουρδικό, είναι ποιος θα κυβερνήσει την Συρία όταν λήξει ο εμφύλιος πόλεμος. Η ευρωπαϊκή διπλωματία και η πολιτική καθώς και η πείρα μας θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν. Έχουμε ζήσει τραγικά γεγονότα εδώ στην Ευρώπη και θα πρέπει να χτίσουμε την ήπια μας δύναμη, την διπλωματία μας, διότι ποτέ δεν θα είμαστε μεγάλη δύναμη από στρατιωτικής απόψεως. Και ένα από τα μέσα είναι και το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, καλωσορίζουμε την Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική και έχει μεγάλη σημασία να την προωθήσουμε όπως κατέδειξαν και τα ε, πρόσφατα γεγονότα στη Βόρειο Αφρική και στη Σαχέλ καθώς και στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να εκπονήσουμε μια τέτοια στρατηγική, αλλά θα πρέπει να, να συζητήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας, ίσως όχι σήμερα, πώς μπορούμε να κινηθούμε στο εγγύς μέλλον. Ποιος είναι ο βασικός μας στόχος για να καταρτήσουμε μία νέα στρατηγική και μέσα στα πλαίσια αυτής της νέας στρατηγικής, ποια είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, δηλαδή τι διαθέτουμε, τι λογισμικό και τι υλικό, τι εξοπλισμό διαθέτουμε μέσα στα πλαίσια και μια συγκεκριμένης πολιτικής θέλησης, διότι συζητήσαμε πραγματιστικά Πολύ χρήσιμη είναι αυτή η συζήτηση, αλλά τι επέρχεται, τι έπεται. Θα πρέπει να θέσουμε επιτάπητος όλες τις ιδέες, στρατηγικές και αρχές που είναι σαφείς για μας, για να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί στους διεθνείς οργανισμούς και φόρα Γιατί αν εκπονήσουμε μια σαφή στρατηγική μπορούμε να είμαστε 27 σε ένα διεθνή οργανισμό, αλλά να μιλάμε με μία φωνή. Τότε δεν τίθεται θέμα. Πρόκειται για την ασφάλεια των πολιτών μας. Πρόκειται για την ασφάλεια και το μέλλον του λόγου και της θέσης μας παγκοσμίω. Εγώ ήμουν υπουργό περιβάλλοντο για δύο χρόνια στη Ρουμανία και ασχολήθηκα με τι κλιματικέ αλλαγέ. Θα πρέπει να το δούμε σαν θέμα ασφάλεια ε, μέσω μακροπρόθεσμα. Ε, Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία να έχουμε ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα, διότι έχουμε εκλογές του χρόνου και ίσως φέτος θα μπορούσαμε να συλλέξουμε αυτά τα ζητήματα για να έχουμε μια εκτενή αλλά συνεκτική στρατηγική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους Υπουργούς ε, για την προκλητική σας εισήγηση αλλά και πολύ σκόπιμα σχόλια. Πολύ μιλήσαμε για την πρόληψη, για την επέμβαση και για την ανοικοδόμηση. Και το θέμα της ευθύνης για προστασία τα συγκαλύπτει όλα αυτά. Θα ήταν σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χτίσει, να ορίσει μία κοινή στάση και συνένεση ως προς την ευθύνη μας για την προστασία των πολιτών μας. Όταν μιλάμε για πρόληψη, για επέμβαση και για νοικοδόμηση θα πρέπει να έχουμε μία διαθεσμική προσέγγιση για να φτάσουμε σε μία ευρωπαϊκή συνένεση. Εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και ίσως αυτό να είναι χρήσιμο και για τα Ηνωμένα Έθνη. Θα ήθελα τις απόψεις σας επ' αυτού. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο υπουργούς για το σχέδιο αυτό, το οποίο είναι αναμενόμενο και το οποίο χρειαζόμαστε ο Καρλ Μπίλτ μίλησε για τις γείτονες χώρες αλλά και τον Ισλαμικό κόσμο που είναι, γιατί πρόκειται για κοντινές χώρες. Ε, μην ξεχνάμε την Τουρκία η οποία δεν προαναφέρθηκε. Νομίζω ότι αν η Τουρκία δεν ήταν υποψήφια χώρα για ένταξη τότε η, τότε η έκθεσή σας του Μαΐου θα ζητούσε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για να ε, γίνει μέλος αλλά έχουν αρχίσει, έχει αρχίσει η προενταξιακή διαδικασία και βρισκόμαστε σε αδίέξοδο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία παγωμένη υποψηφιότητα. Ο Υπουργός Σικόρσκι μίλησε για τις γείτονες χώρες και για το κατά πόσο επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας. Αυτό είναι ένα βασικό θετικό στοιχείο, κάτι το οποίο επιθυμεί η Έφνης η Τουρκία και ε, στοιχεία του Ισλαμικού κόσμου θα ήταν ευπρόσδεκτα στην για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η Τουρκία θα έπρεπε να είναι εντός παρά εκτός. Με την Τουρκία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία θα είναι μέρος της λύσης του προβλήματος. Διαφορετικά αν είναι εκτός θα είναι μέρος του προβλήματος. Συμφωνώ με τον κύριο Σικόρσκι με την περιγραφή του για τις ε, ε, γείτονες χώρες του Νότου. Αλλά πού εντάσσουμε την Τουρκία. Είναι, βρίσκεται νότιο-ανατολικά, ε, βρίσκεται με το ένα πόδι στην Ευρώπη και με το άλλο ε, πέραν του Βοσπόρου, στην άλλη όχθη του Βοσπόρου. Χρειαζόμαστε λοιπόν και το λογισμικό, αλλά το λογισμικό μας και την πολιτική θέληση για να επιλύσουμε το ζήτημα γιατί θα πρέπει να επιληθεί και το θέμα της Τουρκίας κάποια στιγμή, αν όχι στο εγγύς μέλλον, στο απότερο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάπως έτσι, κάπως έτσι είναι. Ε, Jag går Carl kommer förmodligen att protestera min fråga. Det, det har han gjort senaste 20 år då och då. Θα μιλήσω σουηδικά. Τι ίδιες ερωτήσεις κάνω εδώ και 20 χρόνια, αλλά συνεχίζω. Η ερώτησή μου Είναι παραφερή του συναδέλφου. Με ανησυχεί η κατάσταση στον Κάφκασο και δεν βλέπω να βελτιώνεται. Αντιθέτω είναι πιο σοβαρή από ότι εδώ και μερικά χρόνια. Μετά από τα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου, βλέπουμε ότι ίσως θα υπάρξει και συμφωνία σύνδεση με την Αρμενία. Εμείς είπαμε με σαφήνεια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο πριν να υπάρχει βελτίωση στην όλη περιοχή. Η Αρμενία και αποσύρει τα στρατεύματά της. Η Ρωσία δεν ξέρω πώς έχει ενεργήσει. Ποια είναι η απόψή σας. Νομίζω ότι το όλο θέμα και στην περιοχή του Καυκάσου έχει να κάνει και με τη δική μας στάση, όπως και στα Βαλκάν. Και σιγά σιγά το ίδιο θα γίνει. Θα συνεχίσουμε έτσι, θα συνηθίσουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει και κάποια στιγμή θα θεωρήσουμε ότι και με αυτά τα άτομα μπορούμε να συνεργαστούμε, ακόμη και αν δεν ανταποκρίνονται στα δικά μας κριτήρια. Αυτοί λοιπόν μας υποβάλλουν συνέχεια σε αυτή την δοκιμασία. Τι πιστεύετε λοιπόν. Δεν ακούτε καθόλου αυτά που λέμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. <coughs> Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλες δυνατότητες πολιτιστικές, οικονομικές, ε, πνευματικές, οικονομικές και δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι έχουμε να υπομιστούμε και τεράστιες ευθύνες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε κάποια απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις παγκόσμιες, τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, τις σειράξεις διότι είμαστε όλο και πιο ενεργοί σε θέματα επίλυσης διαφορών, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και στην πρόληψη και στην ε, να συγκρότηση μετά από διαφορές. Μίλησαν για το software οι δύο υπουργοί. Όντως, έχουμε το hardware, το οποίο θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί. Και αναφέρθηκε και το επόμενο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε μια μόνιμη θέση στο Συμβούλιο ασφαλεία του ΟΗΕ. Ξέρω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, όλους μα απασχολεί και θα πρέπει να το πολεμήσουμε για να το κατορθώσουμε. Επίση, όταν μιλούμε για το software, δεν θα πρέπει να λιμώζουμε ένα σημαντικό του μέρο. που είναι οι κοινέ αξίε. Ένα από τα συμπεράσματα της ε, Αραβικής Άνοιξης είναι ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει αυτή αυτέ τις, ε, ε, κοινέ αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, να μην τα ξεχνούμε. Ακόμη και στη μερή σχέση μας εκτός Ευρώπης. Ένα από τα συμπεράσματα λοιπόν που συνάγουμε από αυτή την κατάσταση είναι ότι τα οικονομικά συμφέροντα δεν θα πρέπει να δικαιολογούν συνεργασία με καθεστώτα πολιταρχικά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την, ε, την οποία την την όχι μόνο θέτοντας εκείνη στην όλη διαδικασία, αλλά εμβαθύνοντας τη, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και στον πολιτικό και κυρίως πολιτικής και της ασφάλειας. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τις πρωτοβουλίες των δύο Υπουργών τις θεωρώ και ως συμβολή για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο τέλος του χρόνου για τα θέματα άμυνας ε, ε, είναι σημαντικά τα συμπεράσματα από εκεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιοριστούμε στα ε, συνήθιστο στο Συμβούλιο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιήσουμε αυτά που καταφέραμε όλοι μαζί. Ε, η πολιτική γειτονία είναι σημαντική, ε, την αναφέρουν και άλλοι ε, σύμμαχοί μας. Χρειάζεται μια στρατηγική ασφάλειας λοιπόν ενημερωμένη. Υπάρχει εδώ και χρόνια η απόφαση ότι χρειάζεται λευκή βίβλος για την ασφάλεια και την άμυνα όπου θα κάνουμε μια κοινή ανάλυση των απειλών, όπου θα αναφέρεται μια ανάλυση των κοινών μας συμφερόντων, όπου θα διαπιστώνουμε τις συγκεκριμένες μας ικανότητες, μέσα δυνατότητες. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια μιας επανεξέτασης της αμυντικής πολιτικής. Παρακαλώ λοιπόν να συμβάλλετε κι εσείς για, ένα καλό, για καλά συμπεράσματα στο Συμβούλιο και να αποφασιστεί, ε, τουλάχιστον στη, το αργότερο σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, να αποφασιστεί η κατάρτιση Λευκής Βίβλου. Θα μιλήσω πολωνικά. Ε, θα ήθελα ζητήσω από τους υπουργούς να μας πούν τις απόψεις τους σε σχέση με, την, ε, με το δίπολο τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Η Ρωσία δεν θεωρεί ότι υστερεί στο παγκόσμιο στερέωμα. Οι Ρώσοι τώρα χτίζουν ε, το στρατιωτικό τους δυναμικό και σε, άλλες, σε, μετασοβιετικές, ε, σε άλλα μετασοβιετικά κράτη. Και ε, οι κλιματικές αλλαγές αλλάζουν τα δεδομένα Και ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι πλέον η Ρωσία θα έχει πρόσβαση σε νέες ε, πηγές ενέργειας, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Συνεπώς, αυξάνεται ο ρόλος της Ρωσίας στο παγκόσμιο στερέωμα. Δυναμώνει η θέση της ε, Ρωσίας. Εμείς σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ τι αντιπροβάλλουμε. Διότι το ΝΑΤΟ παρακολουθεί τις κλιματικές αλλαγές στο Βορρά. Euh. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τους δύο υπουργούς για την μεγάλη τους διάβγεια, κάτι το οποίο είναι ένα ενθαρρυντικό, άκρος ενθαρρυντικό στοιχείο. Το 83 συμμετείχα στο Κοινοβούλιο και στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, έζησα την κρίση της ε, ε Ιουκοσλαβίας και άκουσα τέτοιους διαυγείς λόγους έναντι της παραλυσίας της Ευρώπης για να αντιδράσει και είδαμε πόσος χρόνος χρειάστηκε για να κινηθούμε. 20 χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όπως είπε και ο κύριος ε, Ντανζόν, δημιουργήσαμε μέσα τα οποία δεν χρησιμοποίησαμε. Η κρίση στο Μάλι έδειξε για άλλη μία φορά ότι κανένα ευρωπαϊκό κράτος, όσο μεγάλο και να είναι, δεν έχει την ικανότητα να προωθήσει μία ε, ε, δράση μέσου βελινεκούς. Μιλάμε για οικονομίες κλίμακας που πρέπει να πραγματοποιήσουμε μέσω στρατιωτικής συνεργασίας. Ένα άλλο σημείο το οποίο θεωρώ ότι είναι σαφές κάτι το κραυγαλαίο είναι ότι οι αρχηγοί ε, κρατών και κυβερνήσεων, ιδιαίτερα των παλαιών μεγάλων κρατών, ε, είναι όμοιροι των, ε, της πρόοδου που θα έπρεπε να επιτευχθεί. Και αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας, τότε φοβάμαι ότι θα είμαστε ένα τεράστιο μουσείο, το οποίο δεν θα έχει επιρροή στον πλανήτη. Θα πρέπει να πείσουμε περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια για συμμετοχή. Βρισκόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τίποτα δεν θα κινηθεί εάν τα εθνικά κοινοβούλια δεν πιστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η μακρά μου πείρα με οδηγεί να πω ότι μετά το τέλος της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς παλινόδησαν τα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ λοιπόν τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, τον κύριο Σικόρσκι, διότι μετά το Δουβλίνο, το Μάρτιο, στη Σύνοδο του Δουβλίνου, μετά από την Κύπρο, θα πρέπει να επιτελεστεί πρόοδος έτσι ώστε να έχουμε μια κριτική κοινοβουλευτική μάζα η οποία να μπορεί να πείσει. Σε αυτό το οικοδόμημα δεν μιλάμε μόνο για τον θεσμικό πυλώνα, αλλά η Αντιπρόεδρος Επιτροπής, η κυρία Άστον, θα πρέπει να ασχοληθεί με πολλά θέματα. Χρειάζεται πολλούς συνεργάτες, έναν για την πολιτική, ένα για το στρατιωτικό σκέλος και επίσης ένας, ο, ο Επίτροπος Ανάπτυξης έχει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ε, ρόλο και χρειάστηκε να μεταβώ στο Αφγανιστάν για να ε, πιστώ από κλιμάκιο του ΝΑΤΟ ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ε, συνεργασία. Υπήρξαν πολλές επιφυλάξεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γιατί υπάρχει και το πολιτισμικό χάσμα μεταξύ του κόσμου της άμυνας και του κόσμου της ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να γεφυρωθούν οι διαφορές. Εάν είχαμε καταφέρει περισσότερα ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια στο Αφγανιστάν, τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα και για το Αφγανιστάν και για τη Βόρεια Αφρική και επειδή η ιστορία στο Μαλί και στο Σαχέλ θα κρατήσει για πολλά χρόνια, ελπίζω οι ευρωπαϊκές χώρες να βοηθήσουν βοηθήσουν εκείνους που πρέπει να διαχειριστούν το πρόβλημά τους. Γιατί ζούμε μία από τις πιο ασταθείς περιόδους για το παρόν και το μέλλον και θα πρέπει να άρουμε αυτή την αστάθεια κατά το δυνατό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε. Η πρωτοβουλία σας είναι πολύ σημαντική. Δεν θα υπάρξει Ευρώπη της άμυνας και ΚΕΠΑ χωρίς να υπάρχει πραγματική κοινή στρατηγική που θα πρέπει να είναι και γραπτή. Νομίζω ότι αυτός είναι απαραίτητος αλλά όχι ικανός όρος για να προχωρήσουν. Μίλησε ο φίλος μας για την ε, εκπρόσωπο. Δεν είναι αυτός ο ρόλος που της ανατέθηκε, για τον οποίο επελέγει. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μία ευρωπαϊκή στρατηγική αν δεν έχουμε πραγματική Ευρώπη. Και καμία Ευρώπη της αν δεν έχουμε Ευρώπη. Δεν θα υπάρχει ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική πριν να έχουμε ένα ομόσπονδο κράτος. Η στρατηγική του Σολάνα του 2003 καλή ήταν στη θεωρία, αλλά ποτέ δεν ε, τέθηκε σε εφαρμογή, διότι πρέπει να τα κατάλληλα μέσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρώπη της άμυνας με μικρά βήματα και με μικρά μέσα, τα οποία δεν θέλει και κανένας να θέσει από κοινού. Να σκεφτούμε τους μεγάλους ε, αεροπορικούς άξονες. Ή, να σκεφτούμε τη συνεργασία μεταξύ Βρετανών και Γάλλων. Η προσέγγιση της Ευρώπης ήταν από πάνω στα κάτω, θα πρέπει να ισχύει το αντίθετο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια Ευρώπη που θα είναι όταν ενεργεί στο Μαλί ή σε άλλες χώρες όταν χρειάζεται. Μπορούμε να έχουμε όλα τα μέσα. Μπορούμε να έχουμε το hardware, το software, τα εργαλεία, τα χέρια και τα πόδια. Αλλά δεν θα πάμε πουθενά αν δεν έχουμε και τον εγκέφαλο, τον ευρωπαϊκό εγκέφαλο που θα είναι σε θέση να σκέπτεται και κυρίως να προωθεί τα συμφέροντα της Ευρώπης. Και να λέμε εμείς οι Ευρωπαίοι και όχι εμείς οι Γάλλοι. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αν έχετε απαντήσεις, ευχαρίστω θα τις ακούσω. Ο κύριος από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Δεν ε, υπάρχει ορισμός για το τι θα είναι η Ευρώπη στο μέλλον. Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα. Ε, μια υπερδύναμη αλλά είπα. Δεύτερον, ένας εταίρος κοντά στη ΣΥΠΑ, οι Πολωνοί το λένε αυτό, Ευρωατλαντική Συμμαχία, που θα βοηθήσει τις ΗΠΑ να παίξουν το ρόλο της υπερδύναμης στα πλαίσια του συνασπισμού των προθύμων. Και τρίτον, ένα μόρφωμα πραγματικά πολύ μερές, με βάση την ε, συνένεση. Πρέπει λοιπόν μετά να δούμε τι ε, θεωρώ ότι θα είναι μια σωστή πολιτική ασφάλειας. Ποιες θα είναι οι επεμβάσεις που διεθνώς γίνονται ανεκτές αλλά ξεπερνούν λίγο την εντολή. Ε, για τη Λιβύη υπάρχει μια συνένεση για την απαγόρευση των πτήσεων. Έγιναν και κάτι παραπάνω και τώρα έγιναν ανεκτά. Και τέλος παρεμβάσεις κατά της δεδηλωμένης ε, αντίδρασης κάποιων, όπως στη Συρία. Πώς θα επιλύσουμε όλα αυτά. Αν πούμε ότι θα δημιουργήσουμε υπερδύναμη, είναι σημαντικό να μπορούμε να παίζουμε τον ρόλο διεθνούς αστυνομίας, να παρεμβαίνουμε παντού, Αφγανιστάν, ε, Ιράκ, ε, Ιράν, ε, Ιράκ, ή ε, να μπορούμε να υλοποιούμε τις πολιτικές που θεωρούμε σημαντικές. και κατανοώ απόλυτα τις ιστορικές εμπειρίες της ε, Πολωνίας με τον μεγάλο εξανατολών γείτονα, αλλά νιώθω μια δυσφορία όταν ακούω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μπλοκ ανταγωνιστικό προς τον μεγάλο αντίπαλο. Δεν το είπατε ε, άμεσα, αλλά το υπενηχθήκατε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό θα ήταν σωστό, ούτε είναι μια πολιτική που μπορεί να συγκεντρώσει τη συνένεση. Ο κ. Άρους Βόλσκι. Συγγνώμη, καθυστέρησα. Γιατί ήμουν κάπου αλλού. Συζητούσαμε το Τζορμπαριτζάν. Έλεγξα τι ελέγχθη, ποιο είπε τι και φαντάζομαι θα μπορούσα να συμφωνήσω με όλους όσους θέλουν κάτι το θετικό για την ΚΕΠΟ μας. Αλλά μεταξύ αυτών που θέλουν, που επιθυμούν, που φροντίζουν, θα πρέπει να συμφωνήσουμε αυτά που λέω. Το πρόβλημα είναι ότι όταν φτάνουμε στην ουσία του προβλήματος, να δούμε τι κάνουμε. Και εγώ ως οικονομολόγος θα πω ότι η ουσία είναι το χρήμα. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι οι κρίσεις αυτές προκάλεψαν πολλαπλά παράπλευρα προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτυχεί συζητήσεις που έχουν γίνει πολλές φορές σε επίπεδο κορυφής. Τα τελευταία 7 χρόνια τι βλέπουμε στον προπολογισμό. Εγώ φωνάζω, δώστε περισσότερα λεφτά για την εξωτερική πολιτική. Το αποτέλεσμα το γνωρίζετε. Ε, μιλώντας ειδικά δεν είναι και τόσο κακά τι έγινε και ξέρετε τι συμβαίνει και με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς δεν είμαστε ε, ακόμη ε, τόσο ευτυχείς. Σε πάση περιπτώσει ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν τα πήγε και πολύ άσχημα η χώρα μου. Αλλά ξέρουμε ότι έγιναν τρομερές περικοπές στη κεφάλαιο 4 που αφορά την εξωτερική πολιτική. Πράγμα το οποίο είναι εντελώς αντίθετο με αυτά τα οποία λέμε να ενισχύσουμε το ρόλο μας και με όλο αυτό το μπλα μπλα που και εγώ έχω κάνει. Εγώ ήμουν υπέρμαχος της συνθήκης Λισαβόνας γιατί υπήρχε αυτό ο περίφημο ε, συντελεστής στην εξωτερική μας πολιτική και είμαστε απογοητευμένοι. Ε, θέτουμε στόχου που δεν είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να του χρησιμοποιήσουμε. Αντώνιο, κύριε Υπουργή, μπορείτε να μου σχολιάσετε το εξή. Πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλους αυτού του στόχου που έχουμε θέσει, που είναι αναμφίβολα η ορθή με τη μείωση των χρηματοδοτικών πόρων. Πώς μπορούμε να έχουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερη Ευρώπη με λιγότερους πόρους. Δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Και τώρα στον κύριο Μπίλτ απευθύνομαι. Την δική σας εξωτερική πολιτική την εκτιμούμε ιδιαίτερα. Κυρίως στην, προς τους ε, γείτονες της Ανατολής. Το ξέρετε. Αλλά θα ήθελα να πω το εξή. Υπάρχει μία συνέπεια μεταξύ των δικών σας φιλοδοξιών ως Ευρωπαϊκή Ένωση και της πολιτικής που κάνετε ως χώρα. Έχετε κάνει τρομερές περικοπές και ένα από τα πρώτα θύματα δεν είναι μόνο η ΚΕΠ. Είσαστε εξαιρετικός μας σύμμαχος, εκτιμούμε τις δράσεις σας καθώς και δράσεις του κ. Κισκόφ που είναι και αυτός και εγώ ανατολικό Αλλά με λιγότερα χρήματα τι κάνουμε. Για τεκμηρικούς λόγους όλοι είμαστε σε δύσκολη θέση. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα στο Νότιο Κάφκασο, στη Γεωργία. Και ίσως η τελευταία μας ελπίδα, Μολδαβία, επίσης δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Χαμένη υπόθεση η Γεωργία, στην Ουκρανία μεγάλα ερωτηματικά και διλήμματα και δεν έχουμε χρήματα, ούτε καν λίγα. Εάν έχουμε λοιπόν χώρες και όπως είπε και κάποιος συνάδελφος δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα λόγια πώς μπορούμε να ενεργήσουμε με την ε, ε, πραγματικότητα. Όταν έχουμε μόνο δύο ελικόπτερα από το Βέλγιο που είναι στο Μαλί. Και είδαμε στην περίπτωση της Λιβύης τις αδυναμίες μας. Και όταν είδαμε με ερωτηματικά τι ακριβώς έχει γίνει και από εμά και από τον ΝΑΤΟ στην κατάσταση του Αφγανιστάν. Όταν βλέπουμε την κατάσταση στη Συρία. Πλήρης παράλυση. Άρχισε η Αραβική Άνοιξη και τώρα ούτε καν τις αρχές που θέλουμε να επιβάλλουμε δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Αδιέξοδο στην ε, Λευκορωσία, η Μολδαβία, στην ε, Αρμενία, πρόβλημα στο Αζερβαϊτζάν που είναι τόσο γεωστρατηγικά ε, δύσκολη, ε, ε, σημαντική χώρα, τι γίνεται. Τι μπορούμε λοιπόν να προσφέρουμε αν δεν έχουμε χρήματα για να κάνουμε αυτές τις πολιτικές που θέλουμε. All from side. Από τη δική μας πλευρά, Καρλ, θα ήθελες να αρχίσεις εσύ. Νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολλά τάχθηκα υπέρ των μεγαλύτερων δαπανών στην έρευνα, στην ανάπτυξη. Άλλοι όμως θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες, άλλες κυβερνήσεις. Και αυτό έγινε στην τελική ε, φάση των διαπραγματεύσεων. Όλοι κινήθηκαν προς τις εγχώριες ανάγκες. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις ε, όρισαν άλλες προτεραιότητες. Όμως, το ότι χρησιμοποιήθηκε μία ε, πρόταση, η απαρχή της λύσης του προβλήματος. Αυτό, αυτό, είναι, αυτό είναι το κλειδί για την επίλυση. Αλλά αν, και, αν διπλασιάσουμε τα κονθήλια της ΕΙΕΔ πάλι δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να δικτυώσουμε την ικανότητά μας Μιλάμε για 40.000 ε, ε, διπλωμάτες, μα δεν μιλάμε για Ευρωπαίους ε, διπλωμάτες, για 40.000 Ευρωπαίους διπλωμάτες, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δημιουργήσουμε ορισμένα κομβικά σημεία όπου θα αναπτυχθούν τα δίκτυα. Ο Ράτη και εγώ, καθώς και μερικοί άλλοι σε άλλα φόρα, Έχουμε ταξιδέψει μαζί, βρεθήκαμε στη Σερβία και στη Μολδαβία με τον William Hague. Ε, όταν διμερώς ε, συζητούμε για τις σχέσεις μας στη Σουηδία με άλλες χώρες και ούτω καθεξής, όλα βαίνουν καλώς. Ψυχολογικά όμως όταν είμαστε 4-5 υπουργοί εξωτερικών, έχουμε κοινά σημεία ε, που μας προβάλλει η ΕΕΔ, αλλά το γεγονός ότι είμαστε τρεις που εκπροσωπούμε την Ευρώπη, αυτό έχει μεγαλύτερη δύναμη. Έχουμε μεγαλύτερη δύναμη πυθούς από το να βρισκόμαστε σε διμερές επίπεδο διαπραγματεύσεων, δηλαδή ο Ράντικ, εγώ και ο Βίλιαμ Χέιγ. Ο Βίλιαμ Χέιγ ε, είναι, έχει και πολύ στεναρό λόγο είναι ε, Βρετανός και αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις. Αυτή είναι η δικτύωση για την οποία σας ε, μίλησα. Αλλά και η συζήτηση έχει μεγάλη σημασία διότι η Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική δεν αφορά μία άσκηση επί χάρτου. Είναι η διαδικασία για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί όπως ε, ξέρετε το πολιτισμικό υπόβαθρο είναι πολύ διαφορετικό στη Σουηδία, στην Ελλάδα και στρατηγικά αυτοί που μέτρησαν περισσότερο ήταν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει πολιτισμική διασπορά και αυτό που έχει σημασία είναι η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων έτσι ώστε ψυχολογικά να έχουμε ένα στρατηγικό τρόπο κοινή σκέψης και τότε θα προβούμε στην δικτύωση ικανοτήτων μας για να εκτελέσουμε αυτή τη στρατηγική. Υποβλήθηκαν και άλλα ερωτήματα. Όταν συζητήσαμε παρεμφερή θέματα. Μίλησα για τη βαλκανική πύρα. Είναι πολύ εύκολο να είμαστε η θεωρητική του θέματος στη, ε, ε, στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε την υπαρκτή κατάσταση. Αυτό αφορούσε και το εγχείρημα της Λιβύης. Εγώ είπα, περιμένετε, μας περιμένει και η Συρία γιατί η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη από τη Λιβύη. Δεν υπάρχει ένας μορφότυπος για όλα που μπορούμε να εφαρμόσουμε παντού. Θα πρέπει να γνωρίζουμε, να είμαστε βαθείς γνώστες μιας κατάστασης γεωγραφικά. Μπορεί να γίνει μια θεωρητική συζήτηση, αλλά δεν υπάρχει ένα ενιαίο υπόδειγμα το οποίο μπορεί να ισχύσει παντού. Ως προς την Τουρκία, συμφωνώ Αναφερθήκαμε και στην περίπτωση της Ισλανδίας που είναι μικρότερης εμβέλειας, αλλά η συμμετοχή της Ισλανδίας και της Τουρκίας είναι κρίσιμη, γιατί δείτε τις εναλλακτικέ. Θα αποσυρθούν, θα κινηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. Εάν η Τουρκία δεν είναι μαζί μας, τότε θα στραφεί εναντίον μας ενδεχομένως κάποια στιγμή και τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Η Ισλανδία δεν είναι τόσο μείζον περίπτωση. Δείτε, τις, η μεγαλύτερη δεν είναι ούτε των ΙΠΑ, ούτε της Δανίας, ούτε της Σουηδίας. Ε, δεν είναι η μεγαλύτερη ούτε των ΙΠΑ. Η Κινέζικη πρεσβεία είναι και η μεγαλύτερη στην Ισλανδία διότι το βλέπουν σαν ένα άνοιγμα προσφορά. Και τότε θα πρέπει και εμείς να αγκυροβολήσουμε κατά κάποιο τρόπο στο βορρά για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς ένα άνοιγμα προς τα εκεί. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσαρτήσουμε και την Ισλανδία και την Τουρκία για διαφορετικούς λόγους. Χαίρομαι που η μία Ευρωβουλευτής ε, μίλησε σουηδικά για την Αρμενία. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομερίες. Μίλησα για την υπερνηστερία, για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Πρόκειται για σειράξεις που δεν έχουν ε, επιληθεί. Ήσασταν εκεί πριν από το Δεκέμβρη και οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών κάνουμε τη διαφορά, διότι συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον Υπουργό Εξωτερικών και είχαμε μεγαλύτερη επίπτωση. Τέλος, ο κύριος Κόβαξ μίλησε για το Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί θα πρέπει να είμαστε μόνιμο μέλος. Ε, το Λονδίνο και το Παρίσι δεν συμφωνούν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Έχω όμως και άλλη μία ανησυχία που είναι πιο κοντά μας. Δείτε τα τελευταία χρόνια. Είχαμε, είχαμε δύο υπουργούς από τη Φιλανδία και το Λουξεμβούργο που ταξίδεψαν ανά τον κόσμο και έδωσαν μάχη για μία έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών να έχουν κοινού στόχους, μία κοινή στοχοθέτηση. Όχι να ζητάμε μία έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί τότε γίνεται διάχυση των δυνάμεών μας. Εάν συμφωνήσουμε με βάση την παρούσα κατάσταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αυτό θα ήταν καλό κάποια στιγμή χρονικά αυτό δεν θα, δεν θα συμβεί αύριο, δεν θα έχουμε έδρα αύριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και θα πείσω το θέμα της Ρωσίας στο Ράντικ. Τι θέλετε να μας αναθέσετε προγολαβικά την ε, πολιτική της Ρωσίας. ασχολήθηκε με κάποια θέματα ο Κάρλα και εγώ με κάποια άλλο. Κύριος Πουλέντς έθεσε το σημαντικό θέμα του πώς μπορούμε το pooling και sharing να δουλέψει στην πράξη. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους λειτουργεί το ΝΑΤΟ που πρέπει να διορθώσουμε εάν θέλουμε να φτιάξουμε τη σωστή μας κοιπία, αλλά και κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να συνάγουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που είναι με τον οποίο αναπτύσσουν τα AWOX, Διότι και εμείς συμμετέχουμε, υπάρχουν ε, οι το ρόλο της περιπολίας, τον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε, στις ε, μανούβρες, αν χρειάζεται να παρέμβουμε. Θα πρέπει να είμαστε παρόντες στην εποπτεία όλων αυτών των λειτουργιών. Τώρα, πώς μπορούμε να δικτυωθούμε, να διασυνδεθούμε μεταξύ τους διπλωματικές μας υπηρεσίες. Τρεις ιδέες έχω περί αυτού. Η πρώτη, Οι συνθήκες μας υποχρεώνουν να εξυπηρετούμε τους πολίτες μας στις προξενικές αρχές. Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε είναι να παρέχουμε ένα κατώτερο επίπεδο υπηρεσιών. Και εάν είμαστε σε θέση να εκπροσωπούμε αλλήλους σε ευρύτερο επίπεδο από ό,τι σήμερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θετικά τις ε, διαφορές μας, αν θέλετε, τις παραδοσιακές. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, είναι πολύ πιο ισχυρές σε κάποια γεωγραφικό μέρος του κόσμου από μας και νομίζω ότι και μας, μας ε, συμφέρει να μας εκπροσωπούν πιο ισχυροί όπου γίνεται. Επίσης, το θέμα των θεωρήσεων και όλο αυτό το σύστημα θα μπορούσε να είναι πιο αποδοτικό και σωστό θα ήτανε να πηγαίνουν σε ένα μόνο μέρος οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν θεωρήσεις, ώστε να μην ανοίγονται παραθυράκια από κάθε προξενική αρχή ε, χωριστά σε κάθε πρωτεύουσα χώρας. Δεύτερον, να είναι σε κοινέ εγκαταστάσεις ενδεχομένως κάποιες πρεσβείες, όπως στην ομάδα του Βίσεγκρατ, στην ε, Σουηδία, σε κάποιες χώρες της Βαλτικής. Δεν σημαίνει από κοινού οι πρεσβείες, αλλά επιτρέπουμε να υπάρχουν κάποιοι χώροι τους οποίους να έχουν πρόσβαση διπλωμάτες μιας άλλης χώρας και όπου είμαστε συμβατοί σε αυτό που κάνουμε αυτό έχει κάποια λογική. Και τρίτο και πιο τολμήρα αν θέλετε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ε, της CIS ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ε, εκπροσωπήσεις και έβρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιες χώρες. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες διπλωμάτες, όντως. Το ίδιο όμως σημαίνει και στην ίδια διπλωματική υπηρεσία της Γερμανίας όπως στην Πολωνία. Οι περισσότεροι υπάλληλοι των διπλωματικών μας υπηρεσιών δεν είναι διπλωμάτες. Είναι υποστηρικτικό και επικουρικό προσωπικό. Εμείς 300-3.500 σε μια μεγάλη πρεσβύλα. 7 από αυτούς είναι, 700 ε, ε, μόνο είναι διπλωμάτες. Και θα μπορούσαμε κάνοντας τη σωστή πολιτική να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα και να έχουμε τους διπλωμάτες στον ίδιο χώρο αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο εάν προσλαμβάνουμε τοπικό ε, επικουρικό προσωπικό. Και αυτό είναι κάτι που θα βελτιώσει και την ασφαλεία μας μεταξύ άλλων. Σκέφτομαι κυρίως τις πρεβίες στις εμπόλεμες ζώνες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουμε στην Καμπούλ το σπίτι της Ευρώπης. Φερρυπίν, όπου το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών μας πηγαίνει στην ασφάλεια. Νομίζω ότι έχουμε 5-6 διπλωμάτες στην Καμπούλ που προστατεύονται από 24 άτομα περίπου. Εάν είχαμε λοιπόν μια κοινή περίμετρο στην οποία θα είχαμε ένα οίκημα στο οποίο ο καθένας θα μπορούσε να χαίρει συνθήκων ασφαλείας θα ήταν κάτι το οποίο πολιτικά θα μας έκανε και πιο ισχυρούς, θα έδινε ένα ισχυρό μήνυμα και θα κάναμε και ε, οικονομίες. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ιδέα μπλοκάρεται από τα μεγάλες χώρες. Διότι παντού ε, λένε ότι θα πρέπει να έχουμε μία περιοχή γιατί πρέπει να πληρώνουμε για τους μικρούς. Έτσι λοιπόν έχουμε διασπάθηση πόρων. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπίσουμε αυτή την αρχή. Στις νέες χώρες να κάνουμε αυτό το περίφημο σπίτι της Ευρώπης. Κάθε δεκαετία δημιουργούνται νέες χώρες. Σκεφτείτε το Σουδάν, το Τιμόρ, αλλά ας κάνουμε αυτά τα περίφημα Europe Houses. Τους 20 της Ευρώπης από κοινού για τους διπλωμάτες μας. Skeptical on to... Επίσης, έχω κάποιους ενδιασμούς για τα θέματα της προσοχής, και ο Καλ σε κάποια θέματα. Στην κυρία Μπράντα Παντό ήταν σχετικά εύκολο να καταλήξουμε σε συνένεση για περιπτώσεις οποίες παραβιάστηκε από κάποιον ηγέτη η ευθύνη για την προστασία. Όταν ο Κατάφη απειλούσε όλη την Πενγκάζη με αφανισμό. Από ηθικής πλευράς αυτό το οποίο έγινε δικαιολογείται. Και από τη στιγμή που πέρασε και στην ε, πράξη ο Ασάντ τώρα στη Συρία θα δικαιολογείται και μία παρέμβαση. Αλλά αυτό δεν το κάναμε διότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα συμμετοχής μας σε μια τέτοια εμπόλεμη κατάσταση στην Αγγής Ανατολή. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Διότι αν αποφασίσουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι πρέπει και να ενεργήσουμε και δεν ξέρω αν έχουμε πάντα την ικανότητα ή το θάρρος να το κάνουμε. Δεν θέλω να πω το εξή ω πρώην μέλος στην Τάνκερ. Σκεφτείτε από νομικής πλευράς τι θα πρέπει να κάνουμε όχι μόνο και μόνο για θέματα ε, προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία κάνουν κάποιοι ηγέτες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν να μπουν σε πόλεμο για να απαλλαγούν από τους ηγέτες τους. Εμείς τι κάνουμε εδώ. Αυτούς τους που μας απειλούν θέλουμε να τους διώξουμε. Αλλά το να κάνουμε κάτι κατά ενός ηγέτη κράτους νομίζω ότι δεν θα ήταν από νομικής πλευράς σωστό. Θα ήταν δύσκολο. Αν το κάνουμε όμως, θα έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ ισχυρό όπλο. Συμφωνώ με τον κύριο Γκάμπλερ απολύτως ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Δεκέμβριο θα πρέπει να έχει μία λευκή βίβλο. Δεν θα πρέπει θα πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά. Να δίνουμε και τι δυνατότητε επιλογών. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία. Ήδη ο Κάρλ είπε ότι θα πρέπει να, σχέση με τη Ρωσία και την κατάσταση να καταλήγουμε σε συμπεράσματα για το τι ακριβώς συμβαίνει σε τακτά Εγώ θα πω το εξή πιο τολμηρό. Εγώ εξέτασα την όλη στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας που είχε συμφωνηθεί στα πλαίσια της Γερμανικής Προεδρίας υπό τον Σρέντερ. με του οποίου τις ιδέες για το τι συμβαίνει με τη Ρωσία δεν μας έβρισκε πάντα σύμφωνος. Το έγγραφό μας είναι εξαιρετικό. Ανθρώπινα δικαιώματα, εξυγχρονισμός. Πολύ σημαντικός ο ρόλος των ΜΚΟ στην ε, Ρωσία. Το πρόβλημα όμως είναι το ίδιο με την σφαιρική στρατηγική της Ευρώπης. Ακόμη και αν έχουμε τις σωστές ιδέες, δεν τις εφαρμόζουμε. Άρα χρειάζεται να είμαστε πιο ρεαλιστικοί και να έχουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη για να θέτουμε σε εφαρμογή τις ιδέες μας. take για δύο λεπτά θα σας απασχολήσω γιατί έχουμε λίγο χρόνο μέχρι τη δεξίωση ως προς τη Λευκή Βίβλο εδώ και χρόνο ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα. Γίνεται λόγος για μία λευκή ε, βίβλο για θέματα άμυνας και πάντα αντιτάσσουμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο γιατί κάτι τέτοιο ε, δεν θα μπορούσε να γίνει από ουσιαστικής πλευρά. Οι Γάλλοι συντάσσουν ένα livre blanc και προσπαθούν να ορίσουν τις στρατηγικές τους φιλοδοξίες. Ίσως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συμβατό. Εγώ θεωρώ ότι η έκθεση Τσεκίνη ήταν ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική πράσινη βίβλος, γιατί μια πράσινη βίβλος χρειάζεται, ε, σε σχέση με την ύπαρξη ε, ενίας αγοράς. Γιατί να ορίσουμε ένα, μια πράσινη βίβλο, διότι δεν είναι δεσμευτική, δεν οριοθετεί, αλλά θεωρεί ε, ο, ως συμπεριληπτικό θετικών στοιχείων ακόμα και μια στρατιωτική επιχείρηση στο Μάλι. Γιατί πολλές φορές η στρατιωτική μας ικανότητα δεν είναι επαρκής. Ίσως ε, θα μπορούσε να ισχύσει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά πόσο θα πρέπει να γίνει μέσω κοινοτικού προπολογισμού. αυτό δεν θα το κρίνει ένας ε, στρατιωτικός αναλυτής. Συνήθως τα χρήματα αυτά διατίθενται σε εθνικό επίπεδο και πολλές φορές η κοινή γνώμη δεν συμφωνεί ούτε και η πολιτική αρχηγή. Αλλά υπάρχει ένα κεφάλαιο στον κοινοτικό προϋπολογισμό που θα μπορούσε να αναθεωρηθεί και αφορά την έρευνα. Μία από τις μεγαλύτερες ε, περικοπές ε, στο προσχέδιο των δημοσιονομικών προοπτικών αφορά την έρευνα. Εάν οι χώρες που τα καταφέρνουν καλά ε, είναι αυτές οι οποίες επενδύουν στην έρευνα και στις επενδύσεις, το ξέρουμε, ισχύει στην ε, Γερμανία, στη Σουηδία και σε άλλες χώρες. Εάν τότε ε, κάνουμε και εκεί κάνουμε περικοπές, τότε δεν θα έχουμε ένα σχετικό, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και για τον ορίζοντα 2020 μιλάμε για εφηρμοσμένη έρευνα στο στρατιωτικό τομέα, στο τομέα της άμυνας. Μιλάμε για μακροχρόνια επένδυση σε, αυτούς, σε αυτό το τομέα που έχει μεγάλη σημασία από στρατηγικής πλευράς και νομίζω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε εσείς σε αυτό το σώμα, να προωθήσετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ και τους τρεις. Ήταν μια πολύ ε, ζωηρή συζήτηση, ζωντανή, που μας οδηγεί μπροστά και για τη διαδικασία επανεξέτασης και για την προετοιμασία του Συμβουλίου των Υπουργών και για ε, τις εργασίες των Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί χρειάζεται εδώ η συνεργασία Εθνικών Κοινοβουλίων και Κυβερνήσεων. Οπότε καλό είναι να επιτελέσουμε πρόοδο εκεί. Θα ήθελα τώρα να σας καλέσω έξω, που έχουμε ένα μικρό μπουφέ είναι το ε, τελευταίο γιατί ε, σε λίγο δεν θα υπάρχουν κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια μπουφέ.